Καλημέρα σας. Αρχίζουμε τις εργασίες μας. Τελευταία συνεδρίαση πρώτων διακοπών. Είχα μια συνεδρίαση συντονιστών όπου συζητήσαμε διάφορα θέματα πήραμε αποφάσεις που αφορούν παραδείγματος χάρη το νόμο των ακτών της, στην Ισπανία στην επόμενη συνάντηση των συντονιστών θα συζητηθεί τι συνέχεια θα δοθεί σε αυτό. Ανακοίνωστε στους συναδέλφους την ανάγκη να αλλάξουμε την ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασής μας το Σεπτέμβριο επειδή ο Επίτροπος Σευκόβιτς προσφέρθηκε να αφήσει τη συνεδρίασή μας. Μετά μελετήσαμε μερικά θέματα που αφορούν την επίσκεψη στην Κύπρο, αναφορά 14, σημείο 14 μάλλον σημερινό, θέμα Nord Stream, η επίσκεψη στην Ουέλβα και η επίσκεψη στην Καμπανία. Προκειμένου να γίνει μια συζήτηση εδώ και μετά να καταλήξουμε σε ψηφοφορία και απόφαση στην επόμενη συνεδρίασή μας. Οι συνέφεις Γκρούνι και Βίλαντ δήλωσαν ότι θα απουσιάζουν για προσωπικούς λόγους. Η συνάδελφος Βαλεάν, η συγγήτρια για το σχέδιο του προπολογισμού, θα απουσιάζει για λόγους υγείας την αντικαθιστά συνάδελφος Νικολάη. Για το σημείο 10, τη αιτήση του συναδέλφου Άγκης αναβάλλεται. Για το σημείο 9, ο φάκελος σχετικά με την έκθεση Παλιαδέλη δεν είναι σωστό και μοιράζεται, μοιράζονται τα σωστά έγγραφα αυτή τη στιγμή. Αυτός που υπέγραψε την αναφορά de θα πάρει το λόγο, θα κάνει μια δήλωση. Έχουμε και τον αναφερόμενο του σημείου 14, του κυρίου Κλάιν. 19 για την εξεταστική αποστολή στην ΟΕΛΒΑ θα εγκριθεί στο τέλος της πρωινής συνεδρίασης τη αιτήση του συναδέλφου Μάγερ, ο οποίος υπέβαλε και δύο τροπολογίες αποδεκτές από τον εισηγητή το απόγευμα θα έχουμε παρόντες πολλούς από τους αναφερόμενους και τοπικές και εθνικές αρχές για τη συζήτηση, για την έκθεση, για την επίσκεψη στη καμπανία. Με, μεταξύ των οποίων και ο Τζοβάνι Ρωμάνο, ε, ο οποίος θα εκπροσωπεί την περιφέρεια, τον συναντήσαμε σε μια άτυπη συνεδρίαση της Επιτροπής μας τον περασμένο μήνα στα πλαίσια των Κροάσεων που είχαμε οργανώσει για την επίσκεψη στην Καμπανία. Θα έχουμε τους ανεφερόμενες των Επιτροπών 17 και 18. 17 και 18. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, θα θεωρήσουμε διπλημένο το σχέδιο αυταμερίσης διάταξης. Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης. 4 Μαΐου και 31 Μαΐου 1 Ιουνίου. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, θεωρούνται εγκεκριμένα τα πρακτικά. Σημείο 6. ψηφοφορίας για τις κατάστασεις προβλέψεων του προπολογισμού τη Ένωση για το οικονομικό έτος 2011. Ο κύριος Γιά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να προτείνω μια ε, τροπολογία στη γνωμοδότησή μας προς την Επιτροπή Προπολογισμών. Ε, σε αυτό το σημείο είμαστε ή δεν πρόσεχα και ήμουν Ωραία. Ε, ε, μια προφορική τροπολογία που έχουμε ήδη στείλει στις ε, πολιτικές ομάδες και έχει σχέση και με το διαμεσολαβητή και έχει συμφωνηθεί και με το διαμεσολαβητή. Στο άρθρο 2 συγκεκριμένα το κείμενο λέγει τώρα. Διαπιστώνει ότι η αύξηση των πόρων για το 2011 που ζητάει ο διαμεσολαβητής είναι ε, συν 5,95% για το 2009 και 7,14% για το 2010. Μόλις 0,60% ε, είναι για το 2011, πολύ μετριοπαθής. Και θα προτείναμε την εξής προσθήκη στο άρθρο 2. Αλλά σε αυτό το διάστημα Οικονομικής και Κοινωνικής Κρίσης το Κοινοβούλιο συστήνει ε, ο διαμεσολαβητής να ε, συμφωνήσει με την πρόταση αυτή και να περιοριστεί ε, όσο γίνεται η αύξηση του προπολογισμού για το επόμενο έτος. Όπως σας είπα, έχει αποσταλεί αυτό το κείμενο στις πολιτικές ομάδες και συμφωνήθηκε και με το διαμεσολαβητή. Παρακαλώ λοιπόν να συμφωνήσετε. Äh, Διαπιστώνετε. σε ένα μάξιμο, μου είπα, σε ένα μήνυμο με εννοούσα. Ε, ζητώ συγγνώμη. Γιατί και εγώ δεν έχω πιει καφέ ακόμα και καταλαβαίνετε. Ε, είπα να περιοριστούν σε ένα ελάχιστο οι δαπάνες ε, ε, και Έκανα λάθος προηγουμένως, σας είπα να περιοριστούν στο μέγιστο οι αυξήσεις. Ένα μικρό σχόλιο παρακαλώ. Θέλουμε να βοηθήσουμε το διαμεσολαβητή να κάνει τη δουλειά του. Εννοείται ότι θέλουμε τα χρήματα να ξοδεύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά δεν μπορώ να το καταψηφίσω. Δεν νομίζω ότι έχει τη θέση του εδώ. Δεν μ' αρέσει εμένα έτσι αυτό το δασκαλίστικο. Μην αυτό, μην εκείνο. Νικολάη. Η κυρία Νικολάη. Ευχαριστώ. Η σύσταση αυτή είναι φυσιολογική όταν συζητάμε για την χρηστή διαχείριση. Είτε πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε πρόκειται για το διαμεσολαβητή Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα στα πλαίσια του προϋπολογισμού να ξοδεύει και να προσπαθεί να μειώνει τις δαπάνες. Δεν νομίζω ότι προσθέτει τίποτα στην έκθεση εδώ και είναι και προφορική. Allora, possiamo mettere in votazione... Ας ψηφίσουμε την τροπολογία. Ναι, θα παρουσιάσω την έκθεση εκ μέρους τη συναδέρφου που έχει ένα πρόβλημα στην φωνή και δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Όσον αφορά λοιπόν την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητε του Ευρωπαίου Μεσολαβητή, συνέχισε με ιδιαίτερα τρόπο το έργο του διαμεσολαβητή. προσπαθεί να έχει επικοδομητικές σχέσεις με όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενθαρρύνει τους Ευρωπαίους πολίτες να προσφεύγουν για να υποστηρίζουν τα δικαιώματά τους όταν αυτά παραβιάζονται λόγω της κακής διαχείρισης. Το 2009 ήταν μια πολύ θετική χρονιά για τον διαμεσολαβητή. Προχώρησε πιο γρήγορα στην εξέταση των διαφόρων πρόσφυγων και είχε έτσι καλύτερα αποτελέσματα. Για να συνεχίσει τώρα το έργο του διομεσολαβητή, εκτιμάω ότι ο προπολογισμό του για το 2011 θα έπρεπε να φτάσει στα που σημαίνει μια αύξηση 0,70% σε σχέση με τον προπολογισμό που είχε για το 2010. Αν συγκρίνουμε τον ε, προπολογισμό, λοιπόν, δεν είναι τόσο μεγάλη η αύξηση, οπότε σας συστήνω να την εγκρίνετε. Εκτιμάμε όλους ιδιαίτερα στο έργο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Δεν χρειάζεται να σας μιλήσω για όλες του τις δραστηριότητες. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να το κάνω αυτό εδώ τώρα. Πιστεύω όμως ότι ε, με την οικονομική αυτή αύξηση θα μπορέσει να αποκριθεί στις υποχρεώσεις του και να συνεχίσει το έργο του και τα καθήκοντά του. Προτείνω λοιπόν να συστήσουμε και να υπερψηφίσουμε την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ τη συνάδελφο Νικολάη. Ζητώ συγγνώμη για αυτή την αντιστροφή που έγινε. Ο συνάδελφος Γιάρ ζήτησε το λόγο Έπρεπε να του δώσω το λόγο. Έπρεπε να δώσει πρώτα στη συνάδελφο Νικολάη το λόγο. Αλλά δεν είχα προετοιμαστεί για την παρέμβαση του συναδέλφου Γιάρα. Τώρα, για την τροπολογία Γιάρα. Προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή η τροπολογία. Και τροπολογία συνδέφου Βέρτμαν, τεχνική τροπολογία. Έχει σχέση με τη μετάφραση μόνο προς τα γερμανικά. Την ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Ψηφίζουμε την έκθεση υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Το επόμενο σημείο η ετήσια έκθεση 2009 του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Η συνάδελφος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να θυμίσω ότι κάθε χρόνο ο, ο διαμεσολαβητής παρουσιάζει έκθεση πραγμένων της περασμένης χρονιάς και θα ήθελα να τονίσω ότι η έκθεση το 2009 είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι θυμίζω ότι με τη νέα συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το εξή, ο διαμεσολαβητής εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν διορίζεται εξού και η σημασία του δικού μας θεσμικού οργάνου και της Επιτροπής Αναφορών ιδιαίτερα ο Νικηφόρος Διαμαντούρος κατέθεσε την έκθεσή του επισήμω στις 19 Απριλίου του 2010 στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στη δική μας επιτροπή στις 4 Μαΐου. Θα ήθελα να θυμίσω τι είπε ήδη στην πρώτη ανταλλαγή απόψε ότι ε, υπόθηκε ότι είναι καλά δομημένη η έκθεση, επιτρέπει στον αναγνώστη να δει τι καταγγελίες δέχτηκε, γιατί υπάρχει ταξινόμηση σε κατηγορίες, κακή διαχείριση ε, των θεσμικών οργάνων κτλ. Είναι κεφάλαια. Ε, βλέπουμε σημαντική μείωση του αριθμού των καταγγελιών που δέχεται ο διαμεσολαβητής από 3.406 το 2008 πάμε στις 3.098 και ε, από 13 μήνες έχει περιοριστεί στους 9 μήνες ο χρόνος ε, επεξεργασίας. Όλα αυτά τα λέει η έκθεσή του και δεν θα επιμείνω σήμερα εγώ. Ε, από την άλλη νομίζω ότι η αποστολή του Μεσολαβητή θα πρέπει να ειδωθεί από δύο πρίσματα. Πρώτον, το νομικό πρίσμα που είναι ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη καλή διοίκηση από τα θεσμικά όργανα. Θα πρέπει να γίνεται σεβαστό αυτό το ε, δικαίωμα των πολιτών και αυτό είναι βασικό στοιχείο τη δουλειά του διαμεσολαβητή. Βρισκόμαστε τώρα στο μετέχμιο. Ε, στη τη Λισαβόνα έχουμε το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και αυτό το δικαίωμα ε, είναι δικαίωμα που μπορεί να επικαλεστεί ο πολίτη για να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Νομική βάση λοιπόν Λοιπόν που πρέπει να ενισχυθεί. Για να φτάσουμε ε, σε αυτό το στόχο του πλήρου σεβασμού της καλής διοίκησης, ο διαμεσολαβητής που έχει και υποστήριξη από τη νέα νομική βάση ε, θα πρέπει ε, να είναι ανεξάρτητος από τα θεσμικά όργανα και να λειτουργεί με ακαιρεότητα και να ε, υποδεικνύει ε, τις κατάφορες παραβιάσεις ε, του δικαιώματος αυτού. Σας παραπέμπω εδώ στην παράγραφο 19 της εκθεσής μου που ζητώ να ενημερώνεται η Επιτροπή μας για την εξέλιξη των ε, υποθέσεων των οποίων επιλαμβάνεται ο διαμεσολαβητής. Στη συνέχεια, το άλλο πρίσμα πέρα από το νομικό είναι και το ηθικό. Θα πρέπει να δούμε μια κουλτούρα, ένα πολιτισμό, μια νοοτροπία των υπηρεσιών. Αυτά δεν τα λέει η συνθήκη, αλλά ε, διέπουν τη λειτουργία ε, των θεσμικών οργάνων. Και τι χρειάζεται εδώ. Πρώτον, ο διαμεσολαβητής θα πρέπει, όπως εδώ και χρόνια το πράττει, να συνεχίσει να ε, προωθεί τους φιλικούς διακανονισμούς. Και θυμίζω 56% των καταγγελιών έτσι ρυθμίζονται. Στη συνέχεια θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές του για την επικοινωνία, έτσι ώστε Ευρωπαίοι πολίτες να ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τις δράσει και τις διαδικασίε που υπάρχουν για να γίνονται σεβαστά. Έτσι λοιπόν, στην τελευταία αυτή φάση της τοποθετησή μου πρέπει να πω ότι αξιολογούμε πάρα πολύ θετικά την έκθεση. Προσπάθησα να το βάλω και εγώ στη δική μου έκθεση, ωστόσο προφέρω και σε κάποιες συστάσει. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά το δίκτυο των Ευρωπαίων Διαμεσολαβητών, ε, νομίζω θα πρέπει να αναπτυχθεί και σας παραπέμπω στην παράγραφο 21, 22 και 25. Το δίκτυο του Ευρωπαϊκού των Διαμεσολαβητών είναι σημαντικό εργαλείο και επιτρέπει στο διαμεσολαβητή και τα αντίστοιχα όργανα να διασυνδέονται μεταξύ τους για να έχουν καλύτερη ανταλλαγή εκβέλτιση των πρακτικών και ε, εμπειριών. Ε, κατά τη διάρκεια τη συζήτηση με τον κύριο Διαμαντούρο διαπιστώσαμε ότι ο ίδιο δεν λαμβάνει ακριβείς στατιστικές ε, των περιπτώσεων των οποίων επιλαμβάνονται οι εθνικοί διαμεσολαβητές. Για να γίνει όμω καλή λειτουργία των θεσμικών οργάνων πρέπει να επιμείνουμε σε αυτή την επικοινωνία. Βεβαίω διοργανώνονται σεμινάρια, αποστέλλονται newsletters, φόρουμ συζήτηση που επιτρέπουν στου διάφορου πρωταγωνιστές να συνεργάζονται, αλλά το δίκτυο αυτό μπορεί να βελτιωθεί. Με την ενίσχυση των θέσεων του Εθνικού Διαμεσολαβητού με το Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, του Εθνικών Κοινοβουλίων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο ή μπορούμε να βάλουμε και μια δικτυακή πύλη ίντρανετ. Επιπλέον, δεδομένης και της επικαιρότητα, νομίζω ότι έπρεπε να αναφέρουμε την πρωτοβουλία των πολιτών και το ρόλο που θα μπορούσε εκεί να διαδραματίσει ο διαμεσολαβητής στο διοικητικό σκέλος. Επαναλαμβάνω στη διαδικασία, επιμένω πάρα πολύ, στη διαδικασία ε, ε έγκρισης κατά πόσο είναι δεκτές, δηλαδή αποδεκτέ ή όχι, οι ε, αναφορές και οι καταγγελίες. Σα παραπέμπω στο σημείο 16 εδώ. Και ένα τελευταίο. Στην έκθεσή μου πρότεινα στα πλαίσια της αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού να προβλέπονται και χρηματικές αποζημιώσεις σε περίπτωση ιδιαίτερης και παρατεταμένης καθυστέρησης. Είδαμε πόσο σημαντικό είναι αυτό και λεπτό το θέμα, αλλά η παράγραφος αυτή είναι υπό την αίρεση ότι θα στείλουμε και ένα μήνυμα στους πολίτες ότι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες, μπορεί να τους φαίνονται τεράστια τα χρονικά διαστήματα και ενδεχομένω κάποια στιγμή να χρειάζεται μια αποζημίωση. Βέβαια αυτό εύκολο δεν θα είναι δεδομένη και τη συγκυρία. Σταματώ εδώ και περιμένω ερωτήσεις, σχόλια και κριτικά από τους συναδέλφους. Παραμένω στη διάθεσή σας. Θυμίζω το χρονοδιάγραμμα. 6 Σεπτεμβρίου προθεσμία κατάθεση τροπολογιών και η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας για τις 29. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά της. Εξαιρετική δουλειά. Και είναι πολύ σημαντικό όντως να δείξουμε ότι στηρίζουμε τη δουλειά του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Να δείξουμε ότι υπάρχει χρηστή δίκηση. Το χρειαζόμαστε τόσο πολύ, το βλέπουμε και θα το δούμε και αργότερα στις αναφορές, είναι, βοηθάει, βοηθάει πάρα πολύ, γιατί έτσι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα έγγραφα. Στο Δανέζικο Κοινοβούλιο 20 χρόνια ήμουνα και ξέρετε τι έγινε. Πάρα πολύ καλή νομοθεσία, πολύ καλή εφαρμογή στην πράξη. Έχουμε ένα καλό νόμο, πανηγυρίζουμε και ένα χρόνο μετά τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να τον υποστηρίξουμε τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Πολύ καλή δουλειά έχει γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, ε, Συνάδελφε Μπουσουτήλ, να δώσουμε πρώτα το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρία πράγματα που μας αρέσουν πάρα πολύ σε αυτήν την έκθεση και τα είπε και η συγκήτρια στην παρουσίασή της είναι οι εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας που είναι διαφορετικά προβλήματα πολλές φορές. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ καλή περίπτωση, ένας πολύ καλός τρόπος να φτάνουμε στην ουσία του ζητήματος αντί να περνάμε από τη μία περίπτωση στην άλλη ανάλογα με τα στοιχεία που έχουμε. Επίσης, μας αρέσει πολύ και το ότι τα αποτελέσματα και ότι βοηθούμε και εμείς αυτό. Όπως επίσης για την ταχύτητα με την οποία χειριζόμαστε τις υποθέσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι και μας μας βοηθάει όταν η επεξεργασία γίνεται πιο γρήγορα. Τώρα, μια φιλική συμβουλή για την παράγραφο 18 στην οποία αναφερθήκατε. Μιλάτε για οικονομικές αποζημιώσεις ενδεχομένως στην περίπτωση σαφών και βαρετινόμενων καθυστερήσεων. Ίσως να μπει και σαν ε, τμήμα τροποποίησεων στο δημοσιονομικό κανονισμό, όπου λέει πότε και πώς εκτελεί το προπολογισμό. Και όχι το περιεχόμενο. Για να υπάρξει νέο περιεχόμενο στον προπολογισμό, χρειάζεται μια άλλη διαδικασία. Ακόμα και για να δημιουργηθούν πληρωμές για καθυστερημένη πληρωμή μιας συναλλαγής πρέπει να υπάρχει οδηγία για την καθυστερημένη πληρωμή. Οπότε, φιλική συμβουλή, μην έχετε πολλές ελπίδες για το ότι θα περάσει ως τροπολογία το σημείο αυτό στον δημοσιονομικό κανονισμό με την αναθεώρησή του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Grazie, il collega Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την τόσο καλή της δουλειά. Η παρουσίαση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Συμφωνώ μαζί της για το ότι η υπηρεσία του Ευρωπαίου Μεσολαβητή είναι και μια πολύ σημαντική υπηρεσία, αλλά επιπλέον προσφέρει και πολύ καλά αποτελέσματα στους Ευρωπαίους πολίτες. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή μας να στηρίξει την υπηρεσία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Με αυτό τον τρόπο στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον κόσμο, ότι δηλαδή οι προσφυγές τους λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Τρία πράγματα θέλω να πω για την έκθεση. Πρώτον, συμφωνώ με την ε, κυρία όσον αφορά την εφαρμογή των νόμων. Αυτό πρέπει να τονιστεί. Αλλά δεν πρέπει να τονίζουμε μόνο την προσέγγιση βάση αποτελεσμάτων, αλλά να λέμε ότι οι αποφάσεις του διαμεσολαβητή πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να τίθεται σε εφαρμογή και αυτές. Όταν έχουμε δηλαδή κάποια θετική απόφαση υπέρ ενός πολίτη που υπέβαλε αναφορά, να φροντίσουμε να δίνεται συνέχεια στην απόφαση αυτή του διαμεσολαβητή να υπάρχουν οι σωστές αποφάσεις αλλά και οι σωστές δράσεις στη συνέχεια. Τώρα για την ε, πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών. Εδώ συμφωνώ με την εισηγήτρια που λέει ότι ο διαμεσολαβητής εδώ πρέπει να μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο στην ε, διαδικασία η οποία μας επιτρέπει να δεχτούμε ή να μην δεχτούμε μια πρόταση που έρχεται από τους πολίτες. Πρωτοβουλία των πολιτών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό εδώ. Πάντως, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει να μπούμε στο βάθος του ζητήματος αυτού, στα πλαίσια μια συζήτησης η οποία θα γίνει προσεχώς για την πρωτοβουλία αυτή των Ευρωπαίων πολιτών. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να εμπλεχθεί ο διαμεσολαβητής ώστε να βοηθάει στην επιλογή των αποδεκτών ή μη πρωτοβουλειών των πολιτών. Αλλά ποιος θα είναι ο ρόλος της δικιάς μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Δεν θα έπρεπε να είναι η Επιτροπή Αναφορών εκείνη η οποία θα αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Να αποφασίζει δηλαδή για το αποδεκτό ή μη των πρωτοβουλειών των Ευρωπαίων πολιτών. Κατά τη γνώμη μου, εμείς πρέπει με ξεκάθαρο τρόπο να τοποθετηθούμε πάνω σε αυτό πριν ε, ξεκινάμε να εξετάζουμε τις πρωτοβουλίες των Ευρωπαίων πολιτών. Το τελευταίο στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι η οικονομική αντιστάθμιση όταν υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στις διαδικασίες. Καταλαβαίνουμε ότι είναι βέβαια πολύ καλό αυτό όταν ένας πολίτης περιμένει για πάρα πολύ καιρό ε, θα πρέπει να έχει κάποιο αντιστάθμισμα, κάποια αποζημίωση. Αυτό όμως στα πλαίσια των δημοσιονομικών κανονισμών. Δεν πρέπει να το συμπεριλάβουμε εδώ στην τελική έκθεση για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και την συνάδελφο από τη Βουλγαρία και τώρα θα μιλήσω αγγλικά, λέει ο μιλητής. Ένα θέμα το οποίο δείχνει ότι ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Ευρωπαίου Δημοσιολαβητή είναι πολύ θετικά πράγματα και ότι η Επιτροπή μας τα βλέπει με πολύ θετικό βλέμμα είναι και η προβολή. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να δώσουμε μεγαλύτερη προβολή στο έργο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στις χώρες μας. Βλέπετε, είναι ελάχιστα γνωστοί και οι εθνικοί διαμεσολαβητέ και οι ευρωπαίοι διαμεσολαβητέ στι διάφορε χώρε. Τώρα, όπω είπε και ο κύριο Μπουσάτελ, είναι πολύ γρήγορα να πούμε ότι θα πρέπει ο Ευρωπαίο διαμεσολαβητή ε, θα αποφασίζει για το αποδεκτό ή όχι των πρωτοβουλίων του πολίτη. Κατά το παρελθόν, είναι κάτι άλλο το τι έγινε. Το να προκαταλαμβάνουμε τώρα τη συνέχεια, να κάνουμε προβλέψεις για το τι θα γίνει με τις πρωτοβουλίες των Ευρωπαίων πολιτών, αυτό είναι πολύ νωρίς. Ας δούμε μαζί η Επιτροπή Αναφορών με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και στη συνέχεια σε τριμερή διάλογο με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, να δούμε ποια θα είναι η αρχιτεκτονική τελικά για τις πρωτοβουλίες των Ευρωπαίων πολιτών. Και μόνο μετά να δούμε τι ρόλο θα έχει να παίξει σε αυτό ο Ευρωπαίος Διομεσολαβητής. Κατά τα άλλα, συμφωνώ απόλυτα με τις προτάσεις και είμαι πεπισμένος ότι με τη βοήθεια των πολιτικών ομάδων η έκθεση αυτή θα γίνει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μέγερ. Και εγώ Πιστεύω ότι πρόκειται για μια εξαίρετη έκθεση και ότι μπορούμε κάλλιστα να τη δεχτούμε. Κρατήσαμε θέση αποχής πριν όσον αφορά τις ελάχιστες δαπάνες, γιατί ξεκινάμε από την αρχή που λέει ότι το δημοσιονομικό δικαίωμα εφαρμόζεται και σε αυτό το σημείο. Καταλαβαίνω πάντως πάρα πολύ καλά που οι συνάδελφοι σε μια τέτοια δύσκολη οικονομική στιγμή καταθέτουν μια τέτοια τροπολογία. Τώρα ήθελα να πάρω το λόγο για μία πρόταση που συζητήθηκε ήδη. Είναι αυτό το οποίο έθεσε και ο κύριος Μπουσάτιλ. Ότι δηλαδή η υπηρεσία του διαμεσολαβητή θα αποφασίζει για τις πρωτοβουλίες των Ευρωπαίων πολιτών. Προς το παρόν, φύγεται αυτό το θέμα στην έκθεση. Εγώ όμως νομίζω ότι δεν πρέπει να πάρουμε καμία απόφαση. Μόνο το φθινόπωρο πρέπει να αποφασίσουμε, όχι τώρα. Αν αποφασίσουμε τώρα, σκεφτείτε το εξή. Πρώτον, ο διαμεσολαβητής θα παίζει και πρέπει να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα πλαίσια των πρωτοβουλίων του πολίτη. Σε περίπτωση που υπάρχει κακή διαχείριση πρέπει να προσφεύγει στον διαμεσολαβητή κανείς. Οπότε η διαδικασία αυτή σαφώς τι πρωτοβουλίες δηλαδή των Ευρωπαίων πολιτών, σαφώς και θα περιλαμβάνει και τον Ευρωπαίο Δημοσιολαβητή. Τώρα, να αποφασίζει εκείνο για το αποδεκτό ή όχι, αυτό σημαίνει ότι τον υποβάλλουμε σε προσφυγή στο δικαστήριο. Έχει δηλαδή τότε διαφορετικό ρόλο από αυτόν που έχει σήμερα. Εξάλλου, στην ακρόασή του, ο ίδιο απέρριψε αυτό το ρόλο. Δεν θέλει να αναλάβει αυτό το ρόλο που κανονικά είναι των δικαστηριών. Οπότε, δεν πρέπει να λέμε κάτι τέτοιο εδώ. Αντίθετα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τη συνάδελφο Τσαβά. Θα τη δώσω το λόγο πάλι. Συμφωνώ με το προφανές το οποίο αναφέρεται στο έγγραφό σας για την ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία με την Επιτροπή μας να συνδυαστούν οι εργασίες της, Επιτροπή, Επιτροπής μας σε περιπτώσεις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο διαμεσολαβητής. Για το ευρωπαϊκό δίκτυο του για το διαμεσολαβητή είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός οργανισμός που πρέπει να ενισχυθεί και πρέπει να το σκεφτούμε γιατί συχνά οι εθνικοί διαμεσολαβητέ δεν απαντάνε στον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή. Πολλές φορές όμως λείπει το δίκτυο στο εσωτερικό της κάθε χώρα για τον κάθε διαμεσολαβητή. Θα πρέπει να φροντίσουμε να διαρθρωθεί καλύτερα αυτό το δίκτυο. Και συμφωνώ με τους ε, συνδέσμους που εξέφραζαν τον προβληματισμό τους κατά πόσον τη στιγμή που συζητιέται και θα το κάνουμε σε λίγο το έγγραφο για την λαϊκή πρωτοβουλία ή δημοψήφισμα να πούμε εμείς ποια είναι η γνώμη μας δίνοντας ένα συγκεκριμένο ρόλο για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Και τώρα θα ξαναδώσω το λόγο στη συνάδελφο Νεντέλτσεβα για να κλείσουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και με υποδείξεις και με σχόλια και με κριτική. Δεν περίμενα αυτές οι δύο παραγράφους. Μάλλον περίμενα μια αντίδραση σε σχέση με τις δύο αυτές παραγράφους και σας ευχαριστώ για όλα τα σχόλια για το δημοσιονομικό κανονισμό. Επίσης ευχαριστώ και την Κομισιόν. Καταθέστε τροπολογίες για να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος όσον αφορά την πρωτοβουλία των πολιτών συμφωνώ με τον Μπουσουτήλ και τους άλλους καλό θα είναι σε αυτή τη φάση να είμαστε σχετικά φρόνιμοι προσεκτικοί αυτό που εγώ λέω είναι να μην πάει χαμένη η εμπειρία του δημοσιολαβητή και η εμπειρία της Επιτροπής μας και διοικητικά ε, ακρόαση των αναφερομένων, καταγγελίες κλπ. Εγώ ήμουν πιστή στο πνεύμα. Ίσως ξέφυγα κάπου στο γράμμα. Βοηθήστε με να μπούμε σε λεπτομέρειες περισσότερο ως προς το γράμμα. Σας ευχαριστώ για τις τροπολογίες. Προθεσμία 6 Σεπτεμβρίου. Πρόεδρος, ευχαριστούμε τη συνάδελφα Νεντέλτσεβα. 6 Σεπτεμβρίου για τροπολογίες. Θα ψηφιστεί στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Πρέπει να συζητήσουμε όμως τις τροπολογίες. Πρόεδρος, η ημερήσια διάταξη σας είπα επειδή ο Επίτροπος ζήτησε να είναι παρόν στην Επιτροπή θα αλλάξει. Μία από τις αλλαγές και συμφώνησαν οι συντονιστές θα είναι να γίνει συζήτηση των τροπολογιών. Αναβάλλεται λοιπόν η ψηφοφορία της έκθεσης αυτής. Θα ψηφιστεί αργότερα αφού προηγουμένως συζητηθούν οι τροπολογίες. Το επόμενο σημείο, η ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Δημοσιολογητή κατόπιν σχεδίου σύσταση προς την Κομισιόν όσον αφορά την καταγγελία 676 2008. Το λόγο στην εισηγήτρια κυρία Παλιαδέλη. Ελπίζω να μην κάνω άλλα λάθη, να με παρακολουθεί η γραμματεία. Ε, νιώθω μία μηχανία ότι ανέλαβα σε ανύποπτο χρόνο, μου ανατέθηκε σε ανύποπτο χρόνο υποχρέωση να συντάξω μία αναφορά σε, μια, σε ένα μάλλον σπάνιο ε, ε, σε μια σπάνια περίπτωση, σε μια ειδική έκθεση που κατέλθεσε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής προκειμένου να καταθέσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την μια περίπτωση αδιαφορίας από τη μεριά της Επιτροπής, ε, της Κομισιόν, σε ένα ζήτημα που ενέπιπτε στον τομέα της κακής ε, διοίκησης, σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά ε, όργανα. το λέω αυτό γιατί σε ανίποπτο χρόνο επίσης είχα καταθέσει μια ερώτηση σε συνεργασία με τον συνάδελφο μου τον κύριο Κρήτον Αρσένη προς την Επιτροπή που αφορούσε το θέμα για το, με το οποίο ασχολείται η ειδική αυτή έκθεση του διαμεσολαβητή. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Ε, ομολογώ ότι δεν ήταν εύκολο να συνταχθεί αυτή η έκθεση, όχι μόνο γιατί απαιτούσε ειδικέ νομικές διατυπώσεις, αλλά γιατί πραγματικά μπαίνει στην ουσία των ζητημάτων που τέθηκαν και με αφορμή την προηγούμενη ε, έκθεση. Στον, τον Μάρτιο του 2007, μία μη κυβερνητική οργάνωση ζήτησε, πρόσβαση, ε, ζήτησε από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσβαση σε έγγραφα που αφορούσαν ε, συζητήσεις που είχαν γίνει με, κοινωνικούς εταίρους σχετικά με ρήπους αυτοκινήτων στις επιβατικών αυτοκινήτων. οκτώ μήνες αργότερα η Επιτροπή επέτρεψε την πρόσβαση στα έγγραφα, σε σύνολο 19 εγγράφων, σε 15 έγγραφα αρνήθηκε να δώσει τρία έγγραφα τα οποία αφορούσαν αλληλογραφία με την πόρσε, με την αυτογερμανική ε, αυτοκινητοβιομηχανία πόρσε. Ο καταγγέλων, ε, η μη κυβερνητική οργάνωση, προσέφυγε στον διαμεσολαβητή. Ε, το Σεπτέμβριο του 2008 ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής έλεγξε τις τρεις επιστολές και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επιτροπή κακώς είχε απορρίψει την πρόσβαση στις τρεις αυτές επιστολές. συνέταξε λοιπόν ένα μήνα αργότερα τον οκτώβριο του 2008 ένα σχέδιο σύστασης προς την επιτροπή να παραχωρήσει την πρόσβαση στο σύνολο του περιεχομένου των επιστολών ή να εξετάσει το ενδεχόμενο της εν μέρη δημοσιοποίησης του περιεχομένου τους σύμφωνα με το άρθρο 228 της συνθήκης για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής ένωσης η επιτροπή θα έπρεπε να απαντήσει εντός τριών μηνών από τη λήψη του σχεδίου σύστασης σε, αυτήν την, ε, αυτό το κείμενο του διαμεσολαβητή. Τρεις μήνες αργότερα πράγματι, τον, το τέλος Ιανουαρίου του 2009, η Επιτροπή αποφάσ, ε, ζήτησε συνεχής, έξι συνεχείς παρατάσεις αυτής της προθεσμίας. Είχαν λήξει οι τρει μήνες και ζήτησε στις 23 Φεβρουαρίου του 9, στις 26 Μαρτίου του 9, στις 29 Απριλίου του 9, στις 29 Μαΐου του 9 και στις 29 Ιουνίου του 9, εννέα μήνες δηλαδή μετά την έναρξη αυτής της διαδικασίας, συνεχεί παρατάσεις. Με τη λήξη των προθεσμιών και επειδή δεν λάβαινε απάντηση στο σχέδιο σύσταση, ο Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή στις αρχές Ιουλίου του 2009 απίφθηνε επιστολή προς την Επιτροπή ζητώντας να μάθει τι συνέβη εντωμεταξύ, εάν έχουν κάποια στοιχεία. Στις 17 Ιουλίου του 2009 η Επιτροπή απάντησε πως δεν ήταν ακόμη σε θέση να δώσει τεκμηριωμένη απάντηση στο αίτημα προκειμένου να διατεθούν προς έλεγχο οι επιστολές ε, στην μη κυβερνητική οργάνωση λόγω συνεχιζόμενων διαβουλεύσεων της Επιτροπής με την Πόρσε. Τρεις μήνες αργότερα, στις 30 Σεπτεμβρίου του 2009, η Επιτροπή ενημέρωσε τον, τον διαμεσολαβητή ότι <clears throat> πήρε απόφαση να υπάρξει δυνατότητα μερικής πρόσβασης στις εν λόγω επιστολές. Ένα μήνα αργότερα, τον Οκτώβριο, τέλος Οκτωβρίου του 2009, η επιτροπή ενημέρωσε τον διαμεσολαβητή ότι ανέθεσε τη μετάφραση της απόφασης ε, με βάση την οποία ενημέρωνε την πόρσε ότι αποφάσισε να ζητήσει μερικά κείμενα ε, μερική πρόσβαση σε λόγο επιστολές η απόφαση αυτή ε, ανακοινώνει λοιπόν ότι μεταφράζεται η επιστολή ε, τέλος, Οκτωβρίου, τέλος Οκτωβρίου. Τέλος Νοεμβρίου ο Διαμαντούρος ζητάει αντίγραφο της επιστολής αυτής μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου η επιστολή δεν είχε μεταφραστεί ή δεν είχε σταλεί ακόμη στην Πόρσε. Τον ε, τέλος Φεβρουαρίου του 2010 η νέα Επιτροπή πλέον αποφασίζει να δημοσιοποιήσει μερικώς τις επιστολές και κοινοποιεί την απόφαση της αυτή στην Πόρσε. Είχαν περάσει τρεις μήνες από την, ε, ε, πέντε μήνες από τη λήψη της αρχικής απόφασης. Ε, στις 24 ε, Φεβρουαρίου του 2010 ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής δεν είχε ακόμη στοιχεία για το τι συνέβαινε. Γι' αυτό το λόγο συνέταξε την ειδική έκθεση που είναι το αντικείμενο της ε, σημερινής συζήτησης και της αφορμής για την σύνταξη αυτής της εισήγησης που μου ανατέθηκε. Μάρτιο του 2010, συγγνώμη, συγγνώμη η νέα επιτροπή έδωσε πρόσβαση στις επιστολές. Ε, τέλος Μαρτίου του 2010 η Ομιλούσα μαζί με τον συνάδελφο Κρήτον Αρσένη καταθέσαμε γραπτή ερώτηση προς την Επιτροπή με θέμα την αδιαφάνεια στην επικοινωνία της με γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία κατά την προετοιμασία της νομοθεσίας για τους ρήπους των αυτοκινήτων. Είχε βγει ήδη στις εφημερίδες, από γερμανικές νομίζω εφημερίδες κιόλας, το, ε, αυτή η παράληψη από τη μεριά της Επιτροπής να, να δώσει τα έγγραφα προς, ε, στην μη κυβερνητική οργάνωση και από εκεί πήραμε αφορμή ε, με τον συνάδελφο να καταθέσουμε την ερώτηση. Η απάντηση της Επιτροπής στην ερώτησή μας ένα μήνα αργότερα στις 28 Τετάρτου του 2010 είναι πραγματικά απαράδεκτη. Βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλη, μια μεγάλη ε, αμηχανία καθότι η απάντηση ήταν 18 λέξεις και έχω νομίζω μιλήσει σε προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής μας αυτής ε, η οποία στην ουσία δεν απαντάει τίποτα. Με παραπέμπει, μας παραπέμπει σε μία άλλη ερώτηση που είχε γίνει πριν από κάποιον άλλον Ευρωβουλευτή και η οποία είναι εντελώς άσχετη προς το, αντικείμενο της, το περιεχόμενο της δικής μας ερώτησης. Είναι περίεργα τα πράγματα αλλά ε, ε, στο τέλος Απριλίου εγώ είχα ήδη οριστεί εισηγήτρια για αυτή την Επιτροπή, κάτι που δεν το γνώριζε τότε η, ε, καινούργια Επιτροπή. Γι' αυτό μου έστειλε και αυτή τη σύντομη απάντηση. Ε, τον Ιούνιο του 2010, 18 Ιουνίου, η Επιτροπή μου έστειλε δεύτερη επιστολή. Αυτή τη φορά ήταν ιδιαίτερα μακροσκελής και αναλυτική δεν μπορώ παρά να συνδέσω αυτή την αναλυτική ε, επιστολή με το γεγονός ότι είχε ήδη κοινοποιηθεί ότι θα ήμουν εισηγήτρια στην ειδική έκθεση του διαμεσολαβητή και με αυτή την ε, επιστολή μου ανακοινώνεται ότι, δεν, ε, ότι η Επιτροπή με το να μην απαντήσει εγκαίρως σε τρεις μήνες στον διαμεσολαβητή δεν παραβίασε το άρθρο 228 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή θα διαβάσω το ε, κομμάτι της, ε, τη διατύπωση ακριβώς. Επειδή, το ενδεχόμενο της, επειδή βρισκόταν σε συνεχείς διαβουλεύσεις με την Πόρσε και επειδή η δημοσιοποίηση των, επιστολών πριν να υπάρχει η έγκριση από τη μεριά της Πόρσε θα μπορούσε ενδεχόμενα να οδηγήσει την υπόθεση στα δικαστήρια επειδή ενέπιπτε σε ένα, σε ένα κομμάτι αυτής, ε, του άρθρου ε, του, κανονισμού ε, που προστατεύει τα εμπορικά συμφέροντα ενός τρίτου, του τρίτου, στην περίπτωση αυτή της Πόρσε. Εκτιμώ ωστόσο ότι τα επιχειρήματα που εκτίθενται στο κείμενο της απάντησης προς την ερώτησή μου αυτή δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις της Επιτροπής απέναντι στα λοιπά θεσμικά όργανα. Πιστεύω ότι η Επιτροπή είχε την υποχρέωση με βάση το άρθρο 228 να απαντήσει οπωσδήποτε εντό τριών μηνών στο διαμεσολαβητή. Ακόμη κι αν δεν του δίνει την τελική απάντηση, να του εξηγήσει τι έχει σκοπό να κάνει. Όφιλε δηλαδή να δώσει, ε, ε, ε όφιλε επιπλέον να δώσει ο, η, η ίδια Επιτροπή την ε, δυνατότητα στην Πόρσε, μια προθεσμία, να επιβάλλει στην Πόρσε μια προθεσμία, προκειμένου και η ίδια η Πόρσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και η Επιτροπή στις δικές της, με βάση τον ίδιο μηχανισμό, τον κανονισμό 1049 ε, του 2001. Εκτιμώ επομένως συμπεραίνως ότι παρά την προσπάθειά της να αποδείξει το αντίθετο η Επιτροπή με την επιστολή που μου, ε, έστειλε ε, δηλώνει ότι στην ουσία αγνόησε την υποχρέωση της απέναντι στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή στάση που εκτιμώ πως κάθε άλλο παρά συμβάλλει στο διαθεσμικό διάλογο αλλά και στη θετική δημόσια εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτιμώ αντίθετα πως ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε το όλο ζήτημα κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη συγκεκριμένη περίπτωση τη μη κυβερνητική οργάνωση προς την επιτροπή και αποδυναμώνει τους του τον θεσμό του ευρωπαίου μεσολαβητή και εμέσως επειδή είμαι μέλος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου ε, το ίδιο το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Ε, ζητούμε από την ευρωπαϊκή επιτροπή με την, με την εισήγησή μας αυτή να αναγνωρίσει ότι οι υπερβολικές και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις της στην απάντηση που όφιλε στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή συνιστούν σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση παράβαση του καθήκοντός της για καλόπιστη συνεργασία με τον κύριο Διαμαντούρο. Προσβλέπουμε σε μια δέσμευση της Επιτροπής προς, τον Ευρω... προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα τηρεί την υποχρέωσή της να συνεργάζεται καλή την πίστη με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Και εκτιμούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει αυτή την, δυνατότητα να επιβάλλει αυτή την άποψη ε, δηλώνοντας ότι ε, αν δεν αναλάβει αυτή τη δέσμευση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξακολουθήσει να μην συνεργάζεται με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, το Κοινοβούλιο μπορεί να προχωρήσει σε επιβολή κυρώσεων, ανάμεσα στις οποίες μία είναι και η εγγραφή μέρους του προϋπολογισμού της ε, Επιτροπής για διοικητικές δαπάνες στο αποθηματικό. Η εισήγηση αυτή είχε ένα και μοναδικό στόχο. Να προστατέψει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και να διαφυλάξει το κύρος τους ως προϋπόθεση για την αναβάθμιση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανά της. Η Επιτροπή ως εκτελεστική εξουσία έχει τη μέγιστη υποχρέωση προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν μπορεί να παραπονείται για το κενό, για, το χάσμα ανάμεσα στους πολίτες και την Ευρώπη όταν δεν είναι η ίδια απολύτως συνεπής με τις τυπικές της υποχρεώσεις. Οφείλει, πιστεύω, να σέβεται πρώτη αυτή τη προθεσμία και να αντιμετωπίζει με το δέοντα σεβασμό όχι μόνο τα μέλη του Κοινοβουλίου, όπως η σύντομη απάντηση στην ερώτησή μου, την πρώτη, ερώτηση, ε, η πρώτη σύντομη ε, απάντηση στην ερώτησή μου, αλλά βεβαίω και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Η ειδική έκθεση, αυτή που υπέβαλε ο, ο Διαμαντούρος, είναι το τελευταίο όπλο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή προκειμένου να προασπίσει τη χρηστή διοίκηση στα ευρωπαϊκά όργανα. Και είναι η πρώτη φορά από την ίδρυση του θεσμού το 1995 που γίνεται κάτι τέτοιο, που ο διαμεσολαβητής προσφεύγει στο Κοινοβούλιο για έλλειψη ειλικρινού συνεργασία με κάποια από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω πως η Επιτροπή Αναφορών, η μόνη που βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους Ευρωπαίους πολίτες, και το ομολογούμε όλοι μας αυτό, δεν θα βρεθεί στη δύσκολη θέση που βρέθηκα εγώ να συντάξει και να υποβάλει σχετική έκθεση για ψήφιση στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τη συνάδελφο Παλιαδέλη. Ο κύριος Κλέρκ. Κλέρκ της Κομισιόν. Κλέρκ. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μου δίνει την ευκαιρία να υποστηρίξω τη θέση μας ως ε, μη κυβερνητική οργάνωση φίλη της γης. Θέλω να προσθέσω σε αυτά που είπε η κυρία Παλιαδέλη πριν από λίγο, ότι δηλαδή εδώ δεν πρόκειται για μία περίπτωση. Από τη στιγμή που ε, κατέγραψε την αναφορά στο Κοινοβούλιο ο Ομπούτσμαν. πολλές φορές ε, η Επιτροπή έχει αρνηθεί την πρόσβαση σε έγγραφα σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ε, στην ίδια πάντα βάση. Πολλές φορές οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις πήγανε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστήρια γι' αυτό. Για πάση περιπτώσει, για να επιστρέψω στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο διαμεσολαβητής κατέληξε τον Οκτώβριο 27 Οκτωβρίου του 2008 για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κακώς αρνήθηκε την πρόσβασή μας στα έγγραφα σε επιστολές της Πόρσε. Επίσης είπε δημοσιολαβητής ότι η Κομισιόν έπρεπε να μας δώσει πρόσβαση στις τρεις επιστολές αυτές της ε, Πόρσε, οι οποίες δεν έπρεπε να είναι απόρριτες, έπρεπε να δημοσιοποιηθούν. Όμως για 20 μήνες μετά η Επιτροπή δεν ε, φρόντισε να συμμορφωθεί με αυτά που είπε ο διαμεσολαβητής. Και έτσι δεν ε, συνεργάστηκε με το διαμεσολαβητή, κάτι που αποτελεί παράβαση των υποχρεώσεών της. Η Επιτροπή λοιπόν δεν ε, διαφύλαξε τα συμφέροντα της κοινή γνώμης, αντίθετα της αυτοκινητοβιομηχανίας Porsche. Και επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω τι ακριβώς έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μάλλον τι δεν έκανε. Λοιπόν, για εννέα μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αντέδρασε, όπως είπατε και εσείς, στη σύσταση του Ευρωπαίου Μεσολαβητή. Μόνο τον Ιούλιο του 2009 του έγραψαν λέγοντας ότι έπρεπε ακόμα να έχουν συζητήσεις με την Πόρσε προκειμένου η Πάρσε να συμφωνήσει με τον αποχαρακτηρισμό των γράφων και τη δημοσιοποίησή τους. Χρειάστηκαν 6 μήνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τον Ιανουάριο 11 Ιανουαρίου του 2010 προκειμένου να ενημερώσει την Πόρσε για την πρόθεσή τη να δημοσιοποιήσει τις επιστολές. Δηλαδή λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να ζητήσει τη γνώμη της Πόρσε. Ναι, και τη πήρε έξι μήνες. Στη συνέχεια, μετά την επιστολή αυτή, η Πόρσε κανονικά έχει δέκα μέρες για να αντιταθεί ή για να πάει στα δικαστήρια την ε, Κομισιόν. Όμως, 8 εβδομάδες πέρασαν και η Πόρσε δεν είχε ακόμα αντιδράσει στην επιστολή αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκανε τίποτα, παρόλο που μόνο 10 μέρε χρειαζόντουσαν και μετά μπορούσε να συνεχίσει τη διαδικασία. Δεν το έκανε όμω και δεν δημοσιοποίησε κανένα έγγραφο, δεν μα έδωσε πρόσβαση σε κανένα από αυτέ τι επιστολέ. Ο διαμεσολαβητή πήγε την αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, μόνο όταν έφτασαν τα πράγματα στις εφημερίδες, το Μάρτιο του 2010. Οπότε τότε και η Πόρσα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασαν δημοσιοποιώντας ε, μέρος των επιστολών αυτών, έχοντας όμως διαγράψει κάποια άλλα κομμάτια. Οι φίλοι της γης δηλώνουν ότι είναι προς το συμφέρον της, ε, του κοινού, ενώ ε, το συμφέρον αυτό το παραβίωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή δεν δημοσιοποίησε τις επιστολές. Εμείς ζητούμε όλες οι επιστολές να δημοσιοποιηθούν. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Ευρωπαίος Δημοσιολογητής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κακώς αρνήθηκε την πρόσβαση στο σύνολο των τριών επιστολών πόσε, μια που μόνο μέρος αυτών δημοσιοποίησε. χωρίς επιχειρήματα, μέρος των επιστολών αυτών δεν το δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεν συνέβη αυτό μόνο σε αυτή την περίπτωση. Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Δημοσιολαβητή, και αυτό είναι τι προηγούμενε εβδομάδε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε κακή διαχείριση. Από πλευρά τη Δημοκρατία, λοιπόν, το πιο σημαντικό ζήτημα είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το δημόσιο συμφέρον Δημοσιοποίηση των επιστολών αυτών είναι πιο σημαντικό από τα συμφέροντα μια επιχείρηση σε τόσο γελίο θα έλεγα επίπεδο, η συμπεριφορά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε την εντύπωση και στα μέσα ενημέρωση ότι τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολλά πράγματα να κρύψει και γι' αυτό δεν δημοσιοποιεί ολόκληρε τι επιστολέ Πόρσε. Εμεί πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη αυτή περίπτωση αλλά και η δουλειά του Ευρωπαίου Δημοσιολαβητή και τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών εξυπηρετούνται πολύ καλύτερα εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βάλει το συμφέρον του κοινού στην καρδιά του ζητήματος και πάνω από το συμφέρον μιας εμπορικής επιχείρησης όπως είναι η Πόρσε. Ελπίζουμε να συμμορφωθεί με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί αυτό είναι το συμφέρον του κοινού. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Μάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η διεκπαιρέωση της περίπτωσης αυτής χρειάστηκε πολύ χρόνο. Θα ήθελα όμως να τονίσω ότι η περίπτωση αυτή, όπως είπε και η συγκήτρια στην εισαγωγική της παρατήρησης, ε, η περίπτωση αυτή είναι μεμονωμένη και μοναδική και δεν είναι χαρακτηριστική των σχέσεων Ευρωπαϊκή Επιτροπής Διαμεσολαβητού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη ε, τις παρατηρήσεις του διαμεσολαβητού και θα είδατε ότι στην ετήσια έκθεσή του υπογραμμίζει τις άριστες σχέσεις που διατηρεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ε, έχει μειωθεί ο χρόνο απόκριση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα αιτήματά του. Γιατί χρειάστηκε εδώ τόσο χρόνο αποκλειστικά και μόνο διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε την άδεια της Πόρσε πριν δημοσιοποιήσει την επιστολή και ήθελε να αποφύγει μια κατάσταση διένεξης και περιττής ε, σύγκρουσης. Σύμφωνα με το κανονισμό 1049, όταν τρίτη ζητούν πρόσβαση στα έγγραφα, θα πρέπει να σταθμίσει ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το συμφέρον ε, ε, του ενδιαφερομένου με τα άλλα συμφέροντα. Ε, η ΠΟΣΕ είχε αντιταχθεί στις προτάσεις δημοσιοποίησης για τις τρεις επιστολές επικαλούμενη εμπορικό απόρριτο. Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολούθησε τη διαδικασία διαβουλεύσεων και παραδέχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρειάστηκε πολύ χρόνο γιατί καθυστέρησε πάρα πολύ η εταιρεία Πόρσε. Η χρονολογική περιγραφή δεν είναι τόσο ακριβής όσο ακούσαμε. Δεν χρειάστηκε ένα εξάμεινο για να ρωτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Πόρσε. Αμέσως τη ρώτησε, αλλά παρέμεινε η Πόρσε σιωπήρη για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι γεγονό ότι είχε αποφασίσει το Σεπτέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αγνοήσει τη σιωπή τη Πόρσε και είχε προετοιμάσει μια επιστολή σύμφωνα με τι διαδικασίε που ακολουθεί που ενημέρωνε την εταιρεία ότι θα δημοσίευε την επιστολή και άφηνε στην εταιρεία 10 μέρε, εργάσιμε μέρε, για να προσφύγει ενδεχομένω στα δικαστήρια. Ε, ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέβαλε μια τελευταία, κατέβαλε, συγγνώμη, τελευταία απόπειρα διαλόγου με ε, την Πόρσε για να αποφύγει κάποια νομική διαμάχη που θα καθυστερούσε ακόμα περισσότερο τη δημοσιοποίηση των επιστολών. Και όλες αυτές οι διαδικασίες χρειάστηκαν χρόνο. Η επίσημη επιστολή στην οποία κοινοποιούσε στην Πόρσε ε, την απόφαση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι του μηνό Φεβρουαρίου. Και η Πόρσε αποφάσισε ε, να απαντήσει στις 5 Μαρτίου δεχόμενη τη δημοσιοποίηση. Η επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η ειδική έκθεση περίπου διασταυρώθηκαν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ήταν υπερβολικές όντω οι προθεσμίες στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά παραμένει ε, μεμονωμένη και μοναδική η περίπτωση αυτή και δεν πρόκειται να αναλυφθεί. Στο μεταξύ έχει λάβει μέτρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επιταχύνει τις απαντήσεις προς το διαμεσολαβητή και η αδίποτε καθυστέρηση ε, προσπαθούμε να μην επαναληφθεί το πρόβλημα. Ήταν η πρώτη φορά ε, που ο διαμεσολαβητής ζητούσε ε, να δημοσιοποιεί επιστολές τρίτων με μη σύμφωνη γνώμη μετά από άρνηση ε, του συντάκτη τη επιστολή. Μέχρι τώρα πρόκειται για έγγραφα τη ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι λοιπόν μια πρώτη περίπτωση καινοφανή και που δεν είχε αντιμετωπιστεί στο παρελθόν σε ό,τι αφορά τα όσα περιέγραψε η κυρία Σιγήτρα, θα ήθελα να κάνω την εξή διευκρίνηση. Είναι γεγονό ότι η πρώτη απάντηση ήταν ε, απάντηση επαναπομπή σε, ε, άλλη ε, κοινοβουλευτική ερώτηση. Διαφορετική από εκείνη της ηγητρίας και αυτό οφείλεται σε διοικητικό σφάλμα. Δηλαδή, υπήρξε πρόβλημα μετάφρασης στην αρχική ερώτηση από τα ελληνικά στα αγγλικά και εκείνη ε, που χειρίστηκα την υπόθεση θεώρησαν ότι ήταν ακριβώς η ίδια με την προηγούμενη ερώτηση. Όταν μεταφράστηκε στη συνέχεια σωστά η δεύτερη ερώτηση έγινε συμπληρωματική απάντηση που ήρθε ε, να καλύψει όλα τα προηγούμενα σημεία που είχατε υποβάλει στην γραπτή σας ερώτηση. Και μπορώ να σας διαβεβαίωσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φροντίζει να σέβεται ε, το καθήκον ειλικρινούς ε, συνεργασίας με το διαμεσολαβητή και έχει λάβει και τα αντίστοιχα μέτρα. Σας ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστούμε. Αρχίζει η συζήτηση. Έφνερ. Λοιπόν, Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορώ να σας κρύψω ότι την περίπτωση αυτή τη θεωρώ πραγματικά αφόρητη. Είναι μια διαδικασία που δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να ανεχθούμε και να δεχθούμε. Υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν νόμοι, οδηγίες και κανονισμοί. Και δεν υπάρχουν για να παραβιάζονται, αλλά για να τηρούνται και συγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί είναι προς το συμφέρον των πολιτών. Αλλιώ τι καθόμαστε εδώ και συζητάμε πρόσβαση στα έγγραφα, οδηγίε, κανονισμού, διοργανικέ συμφωνίε για μετά να διαπιστώνουμε ότι εκεί που πραγματικά ε, σοβαρεύουν τα πράγματα δεν τηρούνται οι κανόνε αλλά κολλησιεργούν. Είναι πολύ λεπτή όντω η περίπτωση αυτή. Έχουμε ένα Γερμανό επίτροπο Ζητώ συγγνώμη που το λέω έτσι ως Γερμανός, αλλά θα πρέπει να το πούμε. Γερμανός ο Επίτροπος, γερμανική η αυτοκινητοβιομηχανία και πρόκειται για την προστασία του περιβάλλοντος. Δηλαδή, ο πολίτης στην Ευρώπη και στον πλανήτη και προσπαθεί να επηρεάσει η εταιρεία την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποφύγει μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό το προσπαθούν όλες οι εταιρείες. Οι άλλες επιστολές δημοσιεύονται. Αυτή τη συγκεκριμένη εταιρεία όχι. Το κοιτάει ο δημοσιολαβητής και τι λέει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε εσφαλμένα θα πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα τα έγγραφα και ε, ουδέν αποτέλεσμα. Και τώρα μας λέτε ότι φταίει η μετάφραση και τέτοια πράγματα είναι προφάσεις. Κατά την άποψή μου τελείως απαράδεκτης. Ε, τόση αλληλογραφία ανταλλάχθηκε, πήγαινε έλα. Και τόση ε, φασαρία έγινε και στο διαμεσολαβητή και στην Επιτροπή μας και παντού που ε, αυτή η εξήγηση πραγματικά δεν ευσταθεί σε καμία περίπτωση και δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση και δεν τη δέχομαι με τίποτα. Και σε ό,τι αφορά την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ομολογήσατε και το βρίσκω πάρα πολύ έντιμο ότι δεν πήγαν όλα σωστά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά ταυτόχρονα λέτε ότι είναι μοναδική και δεν ε, είναι αντιπροσωπευτική η περίπτωση αυτή για το τι γίνεται με τα αιτήματα για πληροφόρηση του διαμεσολαβητού. Επιτρέψτε μου τώρα γι' αυτό το λόγο και γι' αυτά που είπατε να παραθέσω την αιτιολογική σκέψη π όπου λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετήρησε μόνο σε τέσσερις από τις 22 περιπτώσεις του 2009 υποθέσεις αυτή την προθεσμία. Στα ελληνικά είναι το ταφ πι λατινικό. Γιατί βάζουμε προθεσμίες αν δεν τις στηρούμε αφού υποχρεούται η εταιρεία να απαντήσει και αρνείται και να απαντήσει και να δώσει τη σύμφωνη γνώμη της και δεν έχει καμία επίπτωση, τίποτα, ούτε καμία δικαιολογία δεν δίνεται. Απλώς λίγη μία προθεσμία, μετά λίγη επόμενη προθεσμία και νέα επιστολή για παράταση προθεσμίας. Ε, τότε γιατί φτιάχνουμε νόμους και κανόνες. Πού θα προσανατολιστούμε, είναι πραγματικά αφόρητη η κατάσταση. Και μπορεί να είναι μοναδική περίπτωση γιατί έχει λάβει αυτή την έκθεση και την έκταση. Αλλά η πρόσβαση στα έγγραφα ε, είναι μια κατάσταση που καθόλου μεμονωμένη πάντα. Βλέπουμε ε, αθέτηση των υποχρεώσεων και των καθηκόντων που απορρέουν από τις συνθήκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Παλιαδέλη. Είναι εξαιρετική η έκθεσή της και πάρα πολύ αντικειμενική και συγκεκριμένη και πολύ ακριβής η παρουσίαση εδώ στην Επιτροπή. Ε, υποστηρίζουμε πλήρως την έκθεση 100% και θα ήθελα μόνο να πω κάτι και στους συναδέλφους στην αιτιολογική σκέψη γιώτα λατινικό λέει ότι ο διαμεσολαβητής κατέληξε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε άδικα ε, την πρόσβαση στα έγγραφα και στο ΕΝ το ΙΔ λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθυστερώντα 15 μήνες αθέτησε την υποχρέωσή τη για συνεργασία με το Δεμεσολαβητή με ειλικρίνεια και καλή την πίστη. Και τέλος, ο διαμεσολαβητής εντόπισε καθυστερήσει σε άλλη μια υπόθεση που σχετιζόταν με την πρόσβαση σε έγγραφα. Ξέρουμε το βιομηχανικό λιμένα στην Τενερίφη εννοεί και σε σχέση με τις ε, υπόλοιπε υποθέσεις, το ΙΣ λέει μόνο σε τέσσερι από τις 22 υποθέσεις αντέδρασε πρόθεσμα. Θα πρέπει να δούμε τα θέματα πολύ πιο ε, προσεκτικά από ό,τι στο παρελθόν και το Κοινοβούλιο να τρίξει και τα δόντια στην Ευρωπαϊκή Τρεπή. Σας ευχαριστώ και για τα όσα είπατε στο τέλος, ε, κυρία Παλιαδέλη, για τις δυνατότητες επιβολής κυρώσεων. Γιατί δεν είμαστε ένας ξεδοντιασμένος τίγρης πλέον. Έχουμε τη δυνατότητα να προβαίνουμε και σε κυρώσεις, αν φαίνεται ότι δεν αντιδρούν ε, όπως θα έπρεπε ενδιαφερόμενοι. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μποστινάρου, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ρυθμίζετε λίγο το χρόνο σας, γιατί έχουμε ακόμα πολλές εκθέσεις να εξετάσουμε και ήδη έχει πάει η ώρα 11.30. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μία πρώτη παρατήρηση. Εδώ δεν συζητάμε θεωρίες και αφηρημένα πράγματα. Μιλάμε για μία συγκεκριμένη παραβίαση των συνθήκων και των ευρωπαϊκών κανόνων που έχουν γίνει αποδεκτοί και θεωρούνται νόμοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μιλάμε για γενικά πράγματα. Δεύτερον, η Πόρσε δεν αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Συνθήκης από όσο ξέρω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος αλλά δεν συνυπογράφει. Για τις δύο λοιπόν παρατηρήσεις. Θα περίμενε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας έρθει με Κάφκα και Ιονέσκο. Γιατί εδώ πρόκειται για το παράλογο. Θέατρο του παραλόγου. Τρίτον. Στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση μπορούμε να δεχτούμε ότι μια εμπορική επιχείρηση, μια πολυεθνική γιατί όχι, να ασκεί τόσο μεγάλη επιρροή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή να δέχεται γι' αυτό να παραβιάσει τις συνθήκες και τις υποχρεώσεις της. Όταν πρόκειται για τις θεσμικές της σχέσεις με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, αυτό είναι πολύ βασικό πώς θα απαντηθεί αυτό το ερώτημα γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε τώρα, αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις γίνεται το ίδιο. Και θα έρθουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, όπου θα υπάρξει κίνδυνος καταστροφής στη θάλασσα, για παράδειγμα, με τα πόβλητα που πετάνε άλλοι στη θάλασσα. Λοιπόν, μπορούμε να βασιστούμε στις απαντήσεις της Επιτροπής. Η Επιτροπή θα συμπεριφερθεί και τότε, όπως συμπεριφέρθηκε τώρα στην περίπτωση της Πόρσε. Οπότε, το συμπέρασμα. Αν το απόρριτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εφαρμόζεται και για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τότε είναι ψευδέστηση να πιστεύουμε ότι ένας κοινό Ευρωπαίος πολίτης είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο θα μπορεί να έχει πρόσβαση και να επωφεληθεί από την διαφάνεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φανταστείτε, Πάλι θεμελιώδες ζήτημα αυτό και ερώτημα. Δεν είναι μια θεωρητική παρατήρηση που γίνεται. Και στο κάτω-κάτω δεν μεταφράστηκε καλά. Μα δεν πρόκειται για μια ιδιωτική επιχείρηση. Η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το μετάφρασε καλά. Καλά αυτό ε, μα σοκάρει. Και προσπαθώ να κρατηθώ έτσι και να είμαι ευγενή. Πώ είναι δυνατόν να δεχτούμε ένα εισηγητής που ορίζεται από την Επιτροπή Αναφορών η ερώτηση να μεταφράζεται λάθος και να έρχεται εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μα λέει «Α, συγγνώμη, ούψ, έκανα λάθος». Μα τι είναι αυτά. Η Britney Spears είμαστε. Τι είναι αυτά. Είναι απαράδεκτο. Και τέλος. Δεν φταίει κανείς. Δεν είναι κανεί υπεύθυνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την κατάσταση ετών παραβίασης των ευρωπαϊκών συνθήκων και για την έλλειψη διαφάνειας. Ένα όνομα. Έχουμε ένα όνομα. Ποιος φταίει. Και δεν είναι τώρα, το λέμε, αστευόμενοι, δώστε με ένα όνομα. Πραγματικά όμως μιλάω. Υπάρχει κανείς που να θεωρείται υπεύθυνο για αυτήν την κακή διαχείριση. Για μένα πρόκειται για μη χρηστή διαχείριση. Τι είναι αυτά, δώστε μας ένα όνομα. Ποιος φταίει, στο κάτω-κάτω να πάει στο δικαστήριο. Όχι θεωρίες. Αλλιώς εσείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορείτε να μας κορυδεύετε συνέχεια, όπως το έχετε κάνει και παλιότερα με το SWIFT. Και πάλι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν εκείνο το οποίο αγωνίστηκε για να στηρίξει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν ήταν το Συμβούλιο ούτε η Επιτροπή. Και πάλι θεμελιώδε ζήτημα κι αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν συνθήκε που καθορίζουν το ρόλο που παίζει το κάθε κοινοτικό έργο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ δεν μπορεί να είμαστε απλώ παρατηρητέ, να καθόμαστε και να κοιτάμε τα πυροτεχνήματα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όποτε εκείνη θέλει. Ευχαριστώ και συγγνώμη αν παρασύρθηκα. Συγχαίρω στον άνθρωπο Μποστινάρο για την ευρεία ε, μουσική γνώση και κουλτούρα που μας επέδειξε ο συνάδελφος Γιάρ. Perfetto il suo Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι, καλά. Λοιπόν, Νομίζω ότι θα πρέπει καταρχάς να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια για τη σαφέστατη έκθεσή της και πολύ καλή έκθεση. Το είπαν όλοι ότι είναι απαράδεκτο αυτό, δεν είναι μεμονωμένη και ε, επεισοδιακή περίπτωση. Ε, επί της αρχής είναι το πρόβλημα για την πρόσβαση στην ενημέρωση και στα έγγραφα. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Τι κατάφερε τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτή την άρνηση. Ακριβώς με αυτή την ανταλλαγή των επιστολών και την αλληλογραφία ήρθε στο επίκεντρο του δημοσίου ενδιαφέροντος. Και τι τη βοηθάει αυτό. Και πολύ ωραία τα λέει η έκθεση. Εγώ έχω ένα πρόβλημα. Με προβληματίζει πραγματικά το εξή. Είναι αρκετά σαφής η έκθεση και αρκετά συνεπής έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να δράσει. Ε, Έχω έτσι λίγο προβληματίζομαι. Με έχει σοκάρει. Είναι και γερμανική εταιρεία. Όταν μια γερμανική επιχείρηση παίρνει μια επιστολή, είναι τελείως φυσιολογικό εντός τεσσάρων εβδομάδων να απαντάει. Ξέρω εγώ, αυτό είναι κοινή πρακτική. Όταν κάποιο σου στέλνει ένα γράμμα με προθεσμία, απαντά εντό τη προθεσμία. Και θέλω η έκθεση πραγματικά να έχει αποτέλεσμα, να κινήσει κάτι. Αυτό είναι το δικό μου πρόβλημα και το Κοινοβούλιο να μπει στο παιχνίδι και ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου κάτι να κάνουμε για να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και την πιστεύω στην κυριολεξία την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι είναι μεμονωμένη περίπτωση, αλλά ακούσαμε προηγουμένω ότι δεν είναι μεμονωμένη. Παραμένουν τα προβλήματα στη διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παίζουν και τι καθυστερήσει. Ε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα όταν έχουμε νόμου, όταν έχουμε κανονισμούς, αυτοί τηρούνται. Χαίρομαι λοιπόν που είναι τόσο σαφής η έκθεση. Έχω μια αφελή ερώτηση. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε όμω για να κινηθούν τα πράγματα. Αλλιώ εκνευριζόμαστε εμεί ε, ε, ακούμε για την κουλτούρα του κυρίου Μποστινάρου που ξέρει και την Britney Spears, αλλά μα ανεβαίνει πίεση και έχουμε κυκλοφορικό πρόβλημα. Η κυρία Παλιαδέλη για να ολοκληρώσει. Συντομία παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όχι, μήπως θα ήθελε η κυρία Μπαμπέσκου πρώτα. Συγγνώμη, είμαι σκιώδη εισηγήτρια από το ΕΛΚ. Δεν μου το είχαν πει, ζητώ συγγνώμη, λέει η πρόεδρο. Μπορώ τώρα. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στην κυρία Παλιαδέλη για την έκθεσή της αυτή. Ως σκιώδης εισηγήτρια από το ΕΛΚ, Βλέπω να μην υπάρχουν ιδιαίτερε διαφορέ ανάμεσα στην πολιτική μα ομάδα και εκείνη και συμφωνούμε με τα όσα αναφέρει το σχέδιο έκθεση. Με απασχολεί και εμένα η περίπτωση αυτή και το γεγονό ότι ο διαμεσολαβητή έφτιαξε ειδική έκθεση λόγω τη έλλειψη συνεργασία από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρόλο που μια μη κυβερνητική οργάνωση ζήτησε κάποια έγγραφη και βάσει του 141 του 2001 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπρεπε να δώσει πρόσβαση αμέσως στα έγγραφα, μόνο πολύ αργότερα έδωσε πρόσβαση σε 15 μόνο επιστολές. Η Πόρσε θεώρησε ότι δεν προστατεύονται τα εμπορικά συμφέροντα της επιχείρησής της εφόσον δημοσιοποιούνταν όλες οι επιστολές. Όμως ο διαμεσολαβητής 27 Οκτωβρίου του 2008 κατέληξε στο ότι κακώς η Επιτροπή δεν έδωσε πρόσβαση στις τρεις τελευταίες επιστολές, όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Ε, παρέτεινε τις προθεσμίες χωρίς να απαντήσει Λέγοντα ότι εξακολουθούσε να είναι σε διαβουλευσει με την τρίτη πλευρά, την Πόρσε δηλαδή. Επίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι έστειλε επιστολή κοινοποίηση στην Πόρσε. Τον Νοέμβριο του 2009 πήρα αντίγραφο τη επιστολή αυτή. Πριν από λίγε μέρε, μαζί με την κυρία Ζέση και την κυρία Γκρούνη, συζητήσαμε με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τον κύριο Διαμαντούρο, ο οποίο επιβεβαίωσε ότι μέχρι τώρα δεν έχει πάρει αντίγραφο της κοινοποίηση που εστάλει στην Πόρσε. Εγώ θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο κάτι τέτοιο. Επίσης, πιστεύουμε, μάλλον η πιστεύουμε ναι, ότι δεν υπήρχε νομική υποχρέωση βάση του 149 να έχει διαβουλεύσεις με την Πόρσε ή η Κομισιόν. Η Κομισιόν από μόνη της αποφάσισε να έχει τέτοιες διαβουλεύσεις. Εμείς αντιλαμβανόμαστε την Κομισιόν που θέλει να τηρεί τους κανόνες, αλλά τότε πρέπει να τηρεί και τις δικές της προθεσμίες. Συμπερασματικά λοιπόν. Εφόσον πήρε 15 μήνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει πρόσβαση στις επιστολές και δεν έδωσε και αντίγραφο της κοινοποίηση στον Όμπουτσμαν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τήρησε τις υποχρεώσεις της για καλή συνεργασία με τον Ευρωπαίδιο Μεσολαβητή είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται εδώ πέρα για κακή διαχείριση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν πρέπει να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ειλικρινά να συνεργάζεται καλά και καλή την πίστη με τον Ευρωπαίο Δημοσιολαβητή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, η Το μικρόφωνο σας. I did not discuss, ε, η προσφυγή προσθέτει κάποια στοιχεία όσον αφορά την ουσία της περίπτωσης αυτής. Εγώ παρέμεινα στην ε, μεταχείριση απονομικής άποψης που επιφύλαξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην περίπτωση αυτή. Και θα παραμείνω σε αυτό. Για να απαντήσω στον κύριο Γιάρη λοιπόν. Πρότεινα στην τελική διατύπωση της έκθεσης αυτής. Να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγνωρίσει ότι τέτοιες καθυστερήσεις δεν πρέπει να επαναληφθούν και να τονίσουμε ότι μεταξύ άλλων μπορούμε να κάνουμε το εξής να παρεύουμε στον προπολογισμό. Τώρα θέλω να πω δύο λόγια στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ. Αυτά που λέτε τα θεωρώ συγγνώμη, απολογία. Αλλά τίποτα επί της ουσίας δεν είπατε. Ξέρω ότι είσαστε σε δύσκολη θέση, ότι δεν είσαστε εσείς προσωπικά υπεύθυνο για όλα αυτά, αλλά πιστεύω ότι τελικά η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή ταπείνωσε όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ή τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για την υπηρεσία του, ταπεινώθηκε και η ίδια. Γιατί αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να ζητήσει να τηρηθούν κάποιες προθεσμίες από μια ιδιωτική επιχείρηση, προκειμένου αυτή να απαντήσει σε ένα ζωτικό ζήτημα, όπως είναι η πρόσβαση ή όχι στις επιστολές αυτές, ε, τότε ταπεινώνεται η οχι στις επιστολες αυτες τοτε ταπεινωνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε κάτι που θα μας βοηθήσει να δείξουμε τη δύναμή μας. Μεγάλη επιτυχία, πρώτο χειροκρότημα. Ένα πολύ ε, θέμα που μας ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ και στην επόμενη συνάντηση την προθεσμία για τις τροπολογίες ε, την έχετε ακούσει 6 Σεπτεμβρίου, όπως και το προηγούμενο κείμενο. Και αν έχουμε χρόνο, θα φροντίσουμε να έχουμε χρόνο να συζητηθούν οι, τροπολογίες, οι τροπολογίες. περάσουμε στο επόμενο σημείο. Το 10 σας είπα, ο Σνέφος Άγκης ζήτησε να αναβληθεί. Οπότε περνάμε στο 11 γνωμοδότηση για τον έλεγχο εφαρμογής του κοινωτικού δικαίου. Είμαι εγώ η συντάκτρια. Αν φέρει στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τον έλεγχο του κοινωτικού δικαίου, κάθε χρόνο υποβάλλεται προς γνωμοδότηση στην Επιτροπή μας. Φέτος ε, το είχαμε κάπως διαφορετικό είναι κατατομής ανάλογα με το αυτά που λέει το παράρτημα. Σε αυτή την ε, τομεακή κατάταξη έχω μια σοβαρή αμέλεια θα έλεγα της Κομισιόν έναντι της ε, εργασίας μας διότι αναφέρονται περιπτώσεις όπως αυτή της Equitable Life όπου πήραμε ενεργό μέρος και η Κομισιόν δεν αναφέρει τίποτα γι' αυτό. Στο έργο μας, στη συμμετοχή μας υπάρχει μια γενική εισαγωγή μικρή στην έκθεση, αλλά αρκετά σημαντική, διότι ορίζει τις διαδικασίες παράβασης και της Επιτροπής Αναφορών μέσα στα πλαίσια του Γενικού Ελέγχου για την τήρηση του κοινοτικού δικαίου που ασκεί η Κομισιόν. Σε αυτή την εισαγωγή η Κομισιόν δίνει πολύ μεγάλο ρόλο στις διαδικασίες παράβασης του κοινοτικού δικαίου σημειώνει με ικανοποίηση του ορισμούς, τις διαδικασίες, το χρονοδιάγραμμα, την επιτυχία στη μείωση του χρόνου χειρισμού και στη συνεπαγόμενη μείωση των, ε, ε των απορρίψεων. Εδώ τώρα βλέπουμε μόνο τη δευτερεύοντα ρόλο των διαδικασιών. Γιατί όπως λέει η ίδια η Κομισιόν στο έγγραφό της, δεν κινούνται πολλές φορές διαδικασίες παράβασης. Κατά λέει η Κομισιόν ότι η Επιτροπή Αναφορών πολύ συχνά αξιολογεί ερωτήσεις και θέματα σχετικά με τη μη σωστή εφαρμογή του κοινωνικού δικαίου με καλά αποτελέσματα ακόμα και αν η Κομισιόν δεν κινεί διαδικασίες παράβασης. Επίσης δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στη μέθοδο που εφαρμόζουμε, στο δημοκρατικό μας ρόλο, που χάρη στην ενεργό συμβολή των πολιτών επιτρέπουν μια συνεχή εποπτεία του που βρίσκεται η εφαρμογή του κοινωτικού δικαίου. Αν η Επιτροπή Αναφορών την πρόσεχε περισσότερο η Κομισιόν στο κείμενό της, θα μπορούσαμε να παίζουμε και ένα ρόλο προληπτικό με πιο άμεσες παραβάσεις πριν γίνει μια παράβαση. Η Επιτροπή μας με τα εργαλεία που διαθέτει και με τη δυνατότητα που έχει να ζητήσουμε να λογοδοτήσουν οι εθνικές και τοπικές αρχές απλοποιεί τις διαδικασίες, μειώνει το χρόνο των τυπικών ανακοινώσεων Όλα αυτά βοηθούν μέσα στο ευρύ πλαίσιο των ελέγχων και της αποδοχής της κοινωτικής νομοθεσίας θα ήταν ακόμα πιο χρήσιμα αν τύχαναν πλήρους εκμετάλλευσης. Η στάση λοιπόν της Κομισιόν δεν είναι και πολύ ανοιχτή έναντι της Επιτροπής μας. Και αυτά επιβεβαιώνεται από την έκθεση αυτή. Αυτή είναι η πρόταση. Μπορούν να γίνουν τροπολογίες. Καλό την Κομισιόν να αναγνωρίσει το ρόλο της Επιτροπής μας και στο ρόλο ελέγχου και εποπτείας της εφαρμογής του κοινωνικού δικαίου να συμμετέχει το Κοινοβούλιο στη διαχείριση του Portal Web κάτι το οποίο έχει ανακοινώσει η Κομισιόν ότι σύντομα θα εισαχθεί ακόμα δεν έχει γίνει βέβαια και συμμετοχή της Επιτροπής μας στη διαδικασία ελέγχου των επιμέρους περιπτώσεων όταν αποτελούν αντικείμενο και αναφοράς. Αυτά είχα να σας πω. Ακούω τα σχόλιά σας. Πρώτα ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, κύριο Στάντλη. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα θέλαμε να πούμε ότι στόχος της έκθεσης μας είναι να παρέχουμε χρήσιμη πληροφόρηση στο Κοινοβούλιο και χαιρόμαστε για τα θετικά ε, σχόλια και το αίτημα να καλύπτουμε ειδικά στην έκθεσή μας και τις αναφορές και εργαζόμαστε πιο σκληρά για να σας δίνουμε την ενημέρωση που επιθυμείτε για ε, συγκεκριμένες και ειδικέ αναφορές που συνδέονται με παράβαση. Ολοκληρώνω αυτό τον καιρό την επόμενη ετήσια έκθεση και προσωπικά συνεργάζομαι ενεργά με συναδέλφους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βεβαιωθούμε ότι την επόμενη φορά θα σας δώσουμε την πληροφόρηση ακριβώς που χρειάζεστε και ζητάτε. Επίσης, έχουμε επαφές μαζί σας ε, για την ιστοσελίδα και τα δικαιώματα των πολιτών που θέλετε να ε, φτιάξετε και με χαρά σας βοηθήσουμε. Επίσης, ε, σε συμφωνία με το Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εξασφαλίσει ότι θα έχετε εγκαίρως ενημερωμένη πληροφόρηση για την ε, πρόοδο των προσφυγών επί παραβάση και των ζητημάτων που ανακύπτουν για να βοηθήσει αυτό το έργο σας στην Επιτροπή σας. Σε ό,τι αφορά το πιλωτικό πρόγραμμα και πώς αυτό γίνεται κάθε φορά. Πρέπει να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αξιολογεί κάθε φορά τις επαφές με τα κράτη-μέλη για τα πιλωτικά προγράμματα και ενημερώνει τους πολίτες ε, για τη δική της αξιολόγηση. Και όπως έχουμε πει και στην έκθεσή μας, πάνω από 40 διαδικασίες προσφυγής επί έχουν ε, προέλθει από πιλωτικά προγράμματα και στη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρακολουθούμε ε, άμεσα με τις υπηρεσίες μας ε, αυτό το θέμα για να γνωρίζουν πάντα οι πολίτες τι χρονή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά τα θέματα. Σε ό,τι φορά τώρα τους συγκεκριμένους αριθμούς ε, θεμάτων που έχουν ε, πρωτοκολληθεί και δεν δίνεται πληροφόρηση, ε, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη πληροφόρηση, πρέπει να σας πω ότι μόλις 10 με 25% των καταγγελιών μπαίνουν στο πιλότο, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί από μόνη της να απαντήσει για τα υπόλοιπα, χωρίς να χρειαστεί να ανατρέξει στα κράτη-μέλη. Εξού και η διαφορά στον αριθμό ε, του όγκου των καταγγελιών που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκείνων που μπαίνουν στο ε, πιλότο. Επίσης, ε, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και δίνουμε ιδιαίτερη μέρημνα στο θέμα της καθυστερημένης μεταφοράς οδηγιών, γιατί αυτό είναι οργανωτικά και μόνο θέματα. σε αντίθεση με την εφαρμογή και υλοποίηση του κοινοτικού δικαίου που είναι πιο περίπλοκο. Αλλά η καθυστερημένη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία μιας οδηγίας είναι απλώς και μόνο θέμα κακής οργάνωσης. Που θα βελτιωθεί αν δοθεί σωστή προσοχή σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά σας. Θα τη στηρίξουμε βέβαια. Μήπως μπορούμε να προσθέσουμε εδώ κάποιες σημαντικές αναφορές. Χρειάζεται τόσο πολύ να υπάρχει μεγαλύτερο σεβασμό στην όλη διαδικασία από την Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ίσως προσπαθήσουμε, αν μπορούμε, να προσθέσουμε κάποια σημεία. Eh, ε, θα υπάρξει χρόνος για τροπολογίες. Όπως πρότεινε και ο Στενεφός Όκεν. Ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Οι απαντήσεις βέβαια ήταν απλώς υποσχέσεις. Θα περιμένουμε. Πάντως θα κάνουμε την έκθεση αυτή. Πάμε στο επόμενο σημείο το 12. Γνωμοδότηση για την πρόταση κανονισμού σχετικά με την πρωτοβουλία των πολιτών. Εισηγητές. Πρώτη η κυρία Γόλης. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνήσαμε, ο Σέφερ και εγώ, ότι εγώ θα σας παρουσιάσω σήμερα την θέση που πρέπει να έχει κυκλοφορήσει σε όλους σας. Είμαστε δύο εισηγητές από την Επιτροπή αυτή και σας διαβεβαιώ ότι η συνεργασία μας πήγε πάρα πολύ καλά και ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη που μας προσέφερε η Γραμματεία. Συνεργαζόμαστε επίσης στενά και με τους δύο εισηγητές στην Επιτροπή Στεγματικών Υποθέσεων, τον κύριο Λαμασούρ και την κυρία Γκουρμάη. Θα επανέλθω σε αυτό αργότερα. Από πλευράς λοιπόν της δικιάς μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, πώς έχουμε προσεγγίσει αυτό το θέμα υπογραμμίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσει καλά αυτό το μέσο πρωτοβουλίας των πολιτών και να είναι όσο γίνεται πιο ανοιχτό και το κοινό να έχει όσο γίνεται πιο εύκολα πρόσβαση σε αυτό. Είναι θέμα ήθους. Δεν μπορούμε να περιορίσουμε την πρόσβαση των πολιτών στο μέσο αυτό. Από την άλλη μεριά, το μέσο αυτό πρέπει να παραμείνει ένα σοβαρό μέσο και να επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν πραγματικά στον καθορισμό της πολιτικής ατζέντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα λοιπόν είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό και αυτή είναι μια πρωτιά τώρα που έχουμε μπροστά μας. Τώρα πώς προσεγγίζουμε αυτό το πράγμα ήταν αυτό το πρώτο σκέλος. Δεύτερον, τι προσπαθώ να λάβω υπόψη μου. Προσπαθώ να λάβω υπόψη μου την τεράστια εμπειρία που έχει η Επιτροπή μας και τα μέλη της όπως επίσης και η γραμματεία της Επιτροπής μας σε διαδικασίες που δεν είναι βέβαια οι ίδιες, γιατί κάθε αναφορά είναι διαφορετική και κάθε αναφορά είναι διαφορετική από μια πρωτοβουλία των ε, πολιτών. Υπάρχουν όμως κοινά σημεία. Ελπίζω τα κοινά αυτά σημεία σε τεχνικό επίπεδο να ληφθούν υπόψη ώστε να καθοριστεί η προσέγγιση της Επιτροπής για το πότε είναι αποδεκτή και πότε όχι μια πρωτοβουλία πολιτών. Αυτή είναι η βάση από την οποία ξεκίνησα. Θα έρθω τώρα πάλι λίγο στη διαδικασία. Πρόκειται για ένα νομοθετικό φάκελο. Δεν ήθιστε η Επιτροπή μας να χειρίζεται τέτοιες υποθέσεις. Είμαστε σε πρώτη ανάγνωση επί του παρόντος. Μπορούμε να πάμε σε δεύτερη ανάγνωση και ακόμα και σε συνδιαλλαγή. Άρα είναι πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ξέρει ποιες είναι οι δυνατότητές του. Βέβαια, κατόπιν τούτου γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι πρόκειται για ένα μέσο που προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας και που έχει τεράστια σημασία για τους πολίτες μας. Οπότε, αν μπορούμε πιο γρήγορα να προχωρήσουμε και να τελειώσουμε με μια πρώτη ανάγνωση, τόσο το καλύτερο. Σίγουρα όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα δικά μας τα δικαιώματα που είναι να φροντίσουμε να καταλήξουμε σε όσο γίνεται καλύτερη λύση και απόφαση. Έχουμε λοιπόν την έκθεση για την Επιτροπή μας αυτή που προετοιμάζεται. Υπάρχει και έκθεση στην Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων. Ελπίζουμε και οι τέσσερις συζητητές μαζί να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε περίπου μία ενιαία έκθεση. Συναντηθήκαμε χτες όλοι μαζί και πρέπει να σας πω ότι είμαι αισιόδοξη μετά από αυτή τη συνάντηση ότι πράγματι θα μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό. Τώρα άπαξ και το φθινόπωρο. Η έκθεση αυτή τελειοποιηθεί και γίνει αποδεκτή από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, τότε βάσει αυτής της έκθεσης μπορούν να ξεκινήσουν ε, τριμερείς διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Όταν δηλαδή οι κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι αρμόδιες έχουν αποφανθεί. Επιτρέψτε μου τώρα να εξετάσω τα κύρια στοιχεία που πιστεύουμε ο κύριος Έφνερ και εγώ ότι είναι σημαντικά για τη συζήτηση. Έχουμε πάντα υπόψη μας ότι έχουμε μία πρόταση της Κομισιόν, ότι κάπου έχει φτάσει σχετικά με αυτή το Συμβούλιο και το ότι υπάρχει ένα έγγραφο εργασίας στην ε, Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων. Η πρώτη καινοτομία θα έλεγα που προσπαθούμε να εισάγουμε είναι όχι τόσο ότι αυτοί οι οποίοι υποβάλλουν πρωτοβουλία πρέπει πρώτα να έχουν πολλές υπογραφές, ίσως 3.000, πριν να προχωρήσει η Κομισιόν στο να θεωρήσει την πρωτοβουλία αποδεκτή όχι. Όχι, κατά τη γνώμη μας. Αυτό δυσκολεύει και δημιουργεί προβλήματα σε έναν σωρό κόσμο. Είναι προτιμότερο η πρωτοβουλία να εγκρίνεται ως αποδεκτή άπαξ και καταγραφή. Όμως, αυτό το οποίο εμεί προτείνουμε είναι προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι πρόκειται για μια σοβαρή πρωτοβουλία και για μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία τη στιγμή της καταγραφής να υπάρχουν κάποιοι από διάφορες χώρες μέλη που να την υποστηρίζουν. Δηλαδή να έχει υπάρξει κάποια διάδραση μεταξύ ανθρώπων σε πανευρωπαϊκή βάση προκειμένου να υποβάλουν μια πρωτοβουλία. Δεν μπορείς δηλαδή να καθίσεις αύριο το πρωί πίνοντας τον καφέ σου online να αποφασίσεις ότι θέλεις να υποβάλεις μια πρωτοβουλία πολιτών. Όχι, πρέπει να την έχεις συζητήσει προηγουμένως σοβαρά με ανθρώπους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για να ζητάμε ένα μεγάλο αριθμό υπογραφών πριν ελεγχθεί το αποδεκτό ή όχι, για μας δεν είναι ρεαλιστικό. Και είναι μεγάλο εμπόδιο για τον κόσμο. Έπειτα, μην ξεχνάτε ότι η Επιτροπή μας και η Γραμματεία μας όλα αυτά τα χρόνια ελέγχει το αποδεκτό των αναφορών χωρίς να έχει κατακλειστεί. Συνεπώς, το ότι λέει η Κομισιόν πως θα κατακλειστεί με πρωτοβουλίες και δεν θα μπορεί να τις χειριστεί και να ελέγξει το αποδεκτό ή όχι, αυτόν πιστεύουμε ότι δεν είναι κάτι ρεαλιστικό. Επίσης πιστεύουμε ότι ο έλεγχος του αποδεκτού ή όχι μιας πρωτοβουλίας πρέπει να είναι κάτι απλό. Συνάδει, έχει τη σωστή μορφή, περιεχόμενο η πρωτοβουλία. Είναι θέμα αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για τα καταπάτηση κάποιας σύμβασης νομοθεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι όλο. Πολύ απλό. Αυτά όσον αφορά το αποδεκτό μιας πρωτοβουλίας. Εμείς προτείνουμε λοιπόν κάτι πιο απλό. Το επόμενο στάδιο τώρα, όπου προτείνουμε κάτι πιο ριζοσπαστικό και απλό, είναι κάτι που απορρέει επίση από την εμπορία που έχουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Έχουμε κάνει διάφορες συζητήσει για το ποιο μπορεί να υπογράψει μια πρωτοβουλία πολιτών και λέμε ότι πρέπει να περιοριζόμαστε σε αυτούς οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου στι ευρωεκλογέ. Εμεί λέμε κάθε πολίτη, κάθε κάτοικο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποβάλει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί λοιπόν, γιατί στο καλό να μην μπορεί η ίδια κατηγορία ανθρώπων να υπογράψει και να συμμετέχει σε μια πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών. Δεν βλέπουμε γιατί να υπάρχει διαφορά. Και ούτε βλέπουμε να πρέπει να υπάρχει πρόβλημα με την ηλικία. Εμείς τους νέους θέλουμε να κάνουμε να συμμετέχουν στο μέλλον της Ευρώπης. Εντάξει, δεν πρόκειται από τα νηπιαγωγεία να μας έρθουν πρωτοβουλίες. Θα έχουμε όμως από νέους. 16 για παράδειγμα ετών και πάνω που θέλουν να συμμετέχουν. Γιατί όχι. Μην τους αποκλείσουμε εφόσον θέλουμε να πετύχει η πρωτοβουλία αυτή. Αυτά προτείνουμε εμείς. Εντάξει, ορισμένοι μπορεί να το βρουν πολύ ριζοσπαστικό, αλλά εμείς θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί και αν θέλουμε η Ευρώπη να είναι πιο κοντά στον πολίτη και οι πολίτες της να συμμετέχουν πιο πολύ στο μέλλον της, αυτό πρέπει να αποφασίσουμε. Θέλουμε επίσης να εγκρίνουμε και μια πλή μεθοδολογία όσον αφορά ε, την υπογραφή. Όνομα και διεύθυνση. Τίποτα άλλο. Δεν θέλουμε να μας δίνουν την ταυτότητά τους, Εντάξει, μπορεί επειδή στη χώρα μα καλώ δεν έχουμε ταυτότητε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμεί θέλουμε να είναι απλή η διαδικασία. Όμω, ξέρουμε ότι σε πολλέ χώρε μέλη πολλοί θα θέλουν κάτι παραπάνω. Και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ελέγχουν τις υπογραφές. Οπότε εμείς θέλουμε να παραμείνει απλή διαδικασία. Τώρα, αν στη διαδικασία θα επιζήσει η πρότασή μας ή τα κράτη-μέλη θα την αλλάξουν, θα δούμε. Πάντως, εμείς, επειδή ακριβώ ως αρχή θέλουμε να κρατήσουμε απλή τη διαδικασία, να προτείνουμε μόνο αυτά τα στοιχεία και τίποτα άλλο. Τέλος, το τελευταίο ίσως, για το οποίο υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, ίσως εξαιτία της εμπειρίας που έχουμε εμείς στην Επιτροπή αυτή. Αν κάποιοι έχουν ε, μπει στον κόπο να κάνουν μια εκστρατεία, να δουλέψουν για να έχουν ένα εκατομμύριο υπογραφές ή παραπάνω για ένα θέμα και το στέλνουν στην Επιτροπή, πρέπει να παίρνουν μια σοβαρή απάντηση. Αυτή η σοβαρή απάντηση, κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να έχει τη μορφή, αρχικά τουλάχιστον, μιας δημόσιας ακρόασης. Τουλάχιστον έλαβα την πρωτοβουλία να μπορούν να συζητήσουν τι ιδέε του με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δημόσια ακρόαση δηλαδή να υπάρχει. Και μετά οι γραπτές απαντήσεις. Και υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η δικιά μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή. Πιστεύω ότι είναι δύσκολο να πούμε πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει πάντα με επίσημο τρόπο να αναμειγνύεται. Μπορεί να υπάρχουν πρωτοβουλίες που υποβάλλονται και με τις οποίες να μην συμφωνεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε να μην θέλουμε να αποφανθούμε σχετικά ή να θέλουμε απλώς να πούμε ότι πιστεύουμε ότι δεν είναι μια καλή ιδέα. Αλλά αυτό μένει πάντα ανοιχτό. Εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα, αν κάτι έρθει σαν νομοθετική πρόταση, να το δούμε. Τη στιγμή που μαζεύονται υπογραφές πρέπει να υπάρχει δυνατότητα βάσει των διαδικασιών που θα ακολουθούμε να μπορούμε είτε να πρωτοστατήσουμε είτε να κάνουμε μια δημόσια κρόαση κατά τη διάρκεια συλλογής υπογραφών. Όπως επίσης να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια δικιά μας ακρόαση με τα άλλα θεσμικά όργανα αφού έχουν συλλεχθεί οι υπογραφές και τότε να αποφασίζουμε ως κοινοβούλιο για μια δικιά μας έκθεση ή ψήφισμα που να ζητάμε νομοθετική δράση συγχρόνως με την πρωτοβουλία των πολιτών. Δηλαδή το Κοινοβούλιο θα πρέπει να μπορεί ανα πάσα στιγμή να διαλέξει τι θα κάνει. Και αυτό θα πρέπει να φαίνεται στην αιτιολογική σκέψη που συνοδεύει την τελική έκθεση. Δηλαδή, άπαξ και υπάρχει κάτι στην νομοθεσία, εμείς να αποφασίζουμε ανάλογα τι θα κάνουμε. Αυτά είναι τα κυρία στοιχεία. Σε αυτή τη βάση έχουμε δουλέψει. Ειλικρινά πρέπει να σας πω ότι όταν συναντηθήκαμε με τους δύο συγητές από την συνταγματική υποτροπή χτες, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες συνένεσης, πολλές δυνατότητες για συνένεση. Και έτσι ξεκινάμε προτείνοντας ένα κείμενο το οποίο θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο. Θα οργανώσουμε και αποκοινούμε τη Συνταγματική Επιτροπή 30 Σεπτεμβρίου κάτι όπου θα συμμετέχουν και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Τώρα, υπάρχει ένα άλλο θέμα στην έκθεσή μας που θέλουμε να υπογραμμίσουμε και αυτό είναι ότι πρέπει να υπάρχει καλή πληροφόρηση και συμβουλές προς τους πολίτες για το πώς μπορούν να προχωρήσουν ε, σε μια πρωτοβουλία πολιτών. Εννοείται ότι η Επιτροπή στην ιστοσελίδα της και σε όλες τις χώρες μέλη πρέπει να υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες, αλλά και από τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διάφορα κράτη-μέλη. Σίγουρα υπάρχει δυνατότητα, και ο κύριος Σέφνερ θα σας τα εξηγήσει, να υπάρχει ένα ανεξάρτητο σώμα που να μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες. Πάντως αυτή τη διαδικασία θέλουμε να την ενθαρρύνουμε, τη διαδικασία δηλαδή πληροφόρησης του πολίτη. Αυτά λοιπόν ήταν τα κύρια στοιχεία όσον αφορά το έγγραφό μας και την διαδικασία που λαμβάνει η χώρα. Πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν μεγάλες προσδοκίες και ότι είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό για αυτούς. Ευχαριστώ. Επειδή δεν έχουμε χρόνο και πολλοί συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο και το κατανοώ. Και αυτά που μας είπε η συνάδελφος Γόλης και ε, στο όνομα των δύο ε, συνεισηγητών και για τους άλλους ε, εισηγητές επιτρέψτε μου να κάνω μια πρόταση σε συνάδελφο Χέφνερ να αφήσει χρόνο για τους αδέρφους να μιλήσουν και να μιλήσει αυτός στο τέλος εξ ονόματος των δύο εισηγητών. Η κυρία Γόλης κάνει την εισαγωγή, ο συνάδελφος Χέφνερ να κάνει το κλείσιμο. Γιατί έχουμε και άλλα τρία σημεία για σήμερα το πρωί και πολλοί συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Ευχαρίστω. Έτσι κι αλλιώς αυτό θα σας πρότεινα κι εγώ. Ακόμα και αν είχαμε συζητηθεί αλλιώ, χρειαζόμαστε χρόνο για τη συζήτηση. Θα πω σύντομα κάτι στο τέλο, αλλά προτιμώ να μιλήσουν πρώτα οι συνάδελφοι. Εξάλλου την έκθεση μαζί την κάναμε και αυτή που, αυτά που είπε η Νταγιάννα με καλύπτουν και εμένα και δεν χρειάζεται να τα συμπληρώσω. Το λόγο λοιπόν καταρχήν στον εκπρόσωπο τη Κομισιόν. Τεντρέρο. Ευχαριστώ. Και εμείς είμαστε εδώ περισσότερο για να ακούσουμε τη συζήτηση παρά για να μιλήσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω έτσι, πολύ ταπεινά και ειλικρινά τους δύο εισηγητές. Το έγγραφο θέσεων αυτό με το έγγραφο προσυζήτηση που έχει συζητηθεί ήδη στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ανοίγει ένα ευρύτατο φάσμα συζητήσεων για διάφορα θέματα Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα που δεν απέχουν πολύ από την τρέχουσα θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Θα τα συζητήσουμε πάντως και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την ευκαιρία να συμμετέχω στη συζήτηση για τη συνέχεια που θα δοθεί. Ευχαριστώ πολύ. Αρχίζει η συζήτηση λοιπόν. Το λόγο έχει ο κύριος Βαλέσα. Καλημέρα σα. θα ήθελα να πω ότι σε ό,τι αφορά το αρχικό έγγραφο, αυτό αφορά κυρίως πολλά οργανωτικά στοιχεία και καθορίζει και τα κριτήρια του αποδεκτού ή μη αποδεκτού της πρωτοβουλίας των πολιτών. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, όλα αυτά καλά και συμφωνώ ότι θα πρέπει να αρκούν για να γνωρίζουμε ότι είναι ένα υπαρκτό φυσικό πρόσωπο και δεν θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διπλής υπογραφής. Σε ό,τι αφορά τώρα τα στοιχεία ταυτότητας, πρέπει να σας πω ότι ο εισηγητής της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων δεν ομιλεί για αυτό το στοιχείο. Νομίζω ότι ενδεχομένως αυτό να διευκολύνει τους πολίτες να ε, προχωρούν ε, στην πρωτοβουλία αυτή. Σε ό,τι αφορά τώρα τα εμπιστευτικά ή απόρριτα στοιχεία, τους αριθμούς ε, ταυτότητας, αυτό είναι αντικίνητρο. Γιατί αν ένας πολίτης δει ότι του ζητούν αριθμό ταυτότητας θα διστάσει να υπογράψει. Και όταν έρθει μετά ένας δημόσιος υπάλληλος και απαιτήσει να αποκαλυφθούν στοιχεία ταυτότητας Και οι υπάλληλοι που το ζητούν αυτό υποτιμούν ε, το πόσο αντικίνητρο είναι. Αφήστε δε που οι πολίτες δεν κυκλοφορούν όλοι με την ταυτότητά τους επάνω του, οπότε δεν μπορεί ε, να γίνεται συλλογή υπογραφών σε δημόσιους χώρους, αν πρέπει κάθε φορά να γράφεις αριθμό ταυτότητας. Ε, η συνέχεια επίσης που δίνεται οι ελεγκτές δεδομένων και ο επόπτης προστασίας προσωπικών δεδομένων λέει ότι όταν έχουμε άλλα στοιχεία στη διάθεσή μας που είναι απαραίτητα για την πρωτοβολία των πολιτών, τότε απαλλάσσεται από την υποχρέωση ε, ο πολίτης να δώσει στοιχεία ταυτότητας. Και πάλι έτσι δεν διευκολύνεται η συλλογή υπογραφών. Παρακαλώ αυτό το θέμα που αφορά τον αριθμό ταυτότητας να διαγραφεί. Και άλλα θέματα πρέπει να συζητήσουμε. Ε, το εύρος ε, της πρωτοβουλίας, το ρόλο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων καθ' όλη τη διάρκεια, γιατί ακόμα δεν είναι καθορισμένος ε, αυτός. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι δεν πρόκειται για αναφορά δεν είναι μια αναφορά που έχει πάρα πολλές ε, υπογραφές πολιτών. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Είναι ένα νέος τρόπος, είναι μια καινοτομία. να ε, γεννιόνται κοινωνικές πρωτοβουλίες στην Ευρώπη ε, μεταξύ των πολιτών για να αυξάνεται η συμμετοχή τους και να συσφίγονται οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους πολίτες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπουσουτήλ. Ευχαριστώ. θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω και τους δύο συγητές για το ενδιαφέρον αυτό έγγραφο εργασίας. Έχω πολλά θέματα να συζητήσω. Πρώτον, σχέσεις ε, με την ΑΦΚΟ. Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Νομίζω θα πρέπει να κάνουμε κοινή συνεδρία οι δύο επιτροπές. Γιατί έτσι εμεί δεν μπορούμε να καταλάβουμε από ποια προοπτική το βλέπουν οι συνάδελφοι της ΑΦΚΟ. Και θα ήταν πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο πάνω κάτω. Κάτι άλλο. Εγώ δεν έχω ε, έγγραφο εργασία ε, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και δεν ξέρω τι συζητούν εκείνοι και κατά πόσο επαναλαμβάνουν στο ίδιο μήκο κύματο με εκείνο που μα έδωσαν η κυρία Γόλη και ο κύριο Χέφνερ. Για τι λεπτομέρειε τώρα του παρόντο εγγράφου θέσεων που το διάβασα και το βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Πρώτον, οι αρχικοί υποστηρικτές, original supporters, καταλαβαίνω τι λέει η κυρία Γόλη, να αποφύγουμε την κατάσταση, ε, να μην έχουμε υπερβολικό αριθμό αρχικών υπογραφών για μια πρωτοβουλία που τελικά δεν θα είναι αποδεκτή και να χάνετε τόση πολλή ενέργεια σε κάτι που πάει χαμένο. Καλώς. Αλλά το να δώσουμε δικαίωμα σε 7 πολίτες από τρει διαφορετικές χώρες να αρχίσουν μια πρωτοβουλία, ε, και αυτό μου, μου φαίνεται ότι πάει ε, στο άλλο άκρο. Σε κάθε αίθουσα των Βρυξελών μπορείς να βρει 7 ανθρώπους από τρία κράτη-μέλη. Τι θα γίνει ξαφνικά όλοι θα μαγειρεύουν μια, μια πρωτοβουλία των πολιτών. Αυτό θέλουμε, νομίζω όχι. χρειάζεται νομίζω μεγαλύτερος αριθμός από τους 7 για να ξεκινάει αυτή η πρωτοβουλία. Να βάλουμε ένα όριο, αλλά όχι τόσο το αντίθετο. Το δεύτερο, το θέμα του αποδεκτού ή μη ε, μιας ε, πρωτοβουλίας. Μπορεί να υπάρχουν παγίδες και πολλά διαφορετικά σημεία. Παράδειγμα, που θα πρέπει να μας ε, απασχολήσουν ενώ θα βάλουμε ένα όριο και να ξέρουν οι πολίτε τι είναι αποδεικτό και τι όχι. Γιατί πολλέ πρωτοβουλίε θα αποδειχθούν ε, στη συνέχεια ενοχλητικές, ε, πολιτικά άστοχε, δύσκολε. Και τι θα τι κάνουμε, θα τις μπλοκάρουμε. Και ποιο θα έχει αυτή την εξουσία. Αν είναι μια πρωτοβουλία πολιτών για μείωση των μισθών, για παράδειγμα, των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υποθέτω αυτό θα πάρει πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές ως πρωτοβουλία. Και εμείς τι θα την κάνουμε. Αυτό είναι αρμοδιότητα δική μας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα τη δεχτούμε την πρωτοβουλία. Θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι για τα ζητήματα αυτά, διότι ακριβώ ο διάβολο κρύβεται στι λεπτομέρειε. Και επίση, αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών Ελπίζω να χρησιμοποιήσω τη σωστή ε, έννοια στα αγγλικά. Ε, θα είναι και ένα στοιχείο που θα μπορεί να καταργεί ε, την ισχύουσα νομοθεσία, την κείμενη νομοθεσία. Δηλαδή θα μπορούν οι πολίτες να ζητούν με πρωτοβουλία τους να καταργηθούν ευρωπαϊκοί νόμοι, να κυρωθούν. Εγώ, για παράδειγμα, θα φανταζόμουν τη βιομηχανία να βρει με χρηματοδότηση ένα τέτοιο τρόπο να ζητάει κατάργηση ε, της ε, ε ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Και το 1979 υπήρξε ένας νόμος κατά του κυνηγιού και θα έρθουν οι κυνηγοί και ξέρω τι σας λέω γιατί είμαι Μαλτέζος και τα γνωρίζω αυτά τα θέματα να ζητούν κατάργηση της νομοθεσίας για την προστασία των πτηνών για να μπορούν να κυνηγούν είμαι υπέρ της πρωτοβουλίας αυτής, αλλά να μην αφήσουμε να ξεφύγει κάθε ελέγχου. Άλλο θέμα. Ε, ε, ισότητα των όπλων. Όταν πρόκειται στην, για τη χρηματοδότηση και την πρόσβαση στους οικονομικούς πόρους, θα πρέπει να υπάρχει ισότητα και όχι να προχωράει μια πρωτοβουλία επειδή κάποιος την υποστηρίζει οικονομικά και μια άλλη που δεν έχει αυτή την οικονομική υποστήριξη ας πούμε της βιομηχανίας να μην μπορεί να προχωρήσει και αυτό είναι ένα άλλο σημείο επίσης ποιοι θα έχουν δικαίωμα να υπογράφουν συμφωνώ απολύτως να είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελεία τελεία δεν μπορεί αυτό να επεκταθεί σε πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν μπορούν να ψηφίζουν για να εκλέγουν ευρωβουλευτές. Δεν μπορούν να έχουν αυτή το δικαίωμα να υπογράφουν την ε, πρωτοβουλία πολιτών. Διότι, όπως ε, υπονοεί και ε, ο τίτλος, είναι η πρωτοβουλία των πολιτών εκείνων που έχουν την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Διότι οι πολίτες μας εκλέγουν και μετά κάνουν νομοθεσία μέσω ημών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς θα μπορούσαμε να φανταστούμε και πρωτοβουλίες όπου η συντριπτική πλειονότητα ε, είναι ε, άνθρωποι που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάλι είναι στρεβλή εκεί η προσώπηση. Τώρα, 18 μήνε για συλλογή υπογραφών, ε όχι, νομίζω είναι υπερβολικό. Πιο λογικό το 12 μήνο, διότι ε, ασκεί και πίεση στου διοργανωτέ να το διεκπαιρεώσουν σωστά, να κερδίσουν μια ορμή, μια κίνηση. 18 μήνε οδηγεί σε αποτελμάτωση. Ε, η εξακρίβωση των υπογραφών είναι πολύ σημαντικό εδώ το θέμα της εμπιστευτικότητα και προστασία των δεδομένων και να έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να διατηρούν κάποια στοιχεία ιδιωτικά τους απόρριτα. Τώρα, κάποιες πρωτοβουλίες που δεν φτάνουν στο 1 εκατομμύριο υπογραφέ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Είναι σαφές ε, ότι χρειάζεται ε, να μπει ένα όριο. Είτε χρειαζόμαστε ένα, ένα εκατομμύριο είτε όχι. Πρέπει να βάλουμε και ένα πύχη. Και τέλος, πώ συμμετέχουν τα θεσμικά όργανα. Θα πρέπει να υπάρξει ρόλος ε, της Επιτροπής Αναφορών εκεί. Έχει τεράστια εμπειρία η Επιτροπή μας ε, στην αντιμετώπιση των πολιτών και θα πρέπει να έχει ένα ρόλο, περιορισμένο ρόλο όμως, σε θέματα αποδεκτού ή όχι της πρωτοβουλίας. Μόνο εκεί να έχουμε λόγο και το λόγο που μας αναλογεί για να δούμε εάν μια πρωτοβουλία που προτείνουν οι πολίτες θα πρέπει να ε, συνεχιστεί ή όχι. Δεν λέγω ότι θα πρέπει να νομοθετούμε για ποιο ρόλο θα πρέπει να έχουμε μετά το στάδιο του αποδεκτού, αν θα το υποστηρίξουμε ή όχι. Όχι, αυτό να το αφήσουμε ανοιχτό. Αλλά όπως είπε και η κυρία Γουόλης, εάν θεωρούμε ότι θέλουμε να προωθήσουμε κάτι, να πούμε ή να μην πούμε τίποτα, αν δεν μας ενδιαφέρει. Και τέλος, ποιος θα δέχεται την τελική πρωτοβουλία, ποιος θα την κάνει δεκτή όταν φτάσει στο τελικό στάδιο. Όπως λέει και η πρόταση, αυτό θα πρέπει να είναι στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη που μακρηγόρησα. con... θα προσπαθήσω ε, να έρθω σε επαφή με ε, τους δύο επόμενους ε, α, μας λένε ότι δεν μπορούν να αναβάλουν τα δύο επόμενα σημεία. Έχει ζητήσει πολλοί κόσμος το λόγο, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Ένα τέταρτο μόλι. Αλλιώς δεν θα προλάβουμε. Παρακαλώ. Η κυρία Λεγκρή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη και να επικεντρωθώ σε άλλα σημεία, να μην επαναλάβω αυτά που είπαν και οι συνάδελφοι. Τόσο καλά, εξάλλου. Πρώτον, η ταυτότητα. Η επαλήθευση στοιχείων ταυτότητας των συνυπογραφών Πιστεύω ότι καλά θα ήταν τις συγκεκριμένες διαδικασίες επαλήθευσης των στοιχείων όσων υπογράφουν την πρωτοβουλία αυτή να μένει στα χέρια των κρατών μελών και να μην είναι στο δικό μας το επίπεδο. Πρέπει τα κράτη-μέλη να εκτιμήσουν πώς θα το κάνουν αυτό. Η κάθε χώρα, ανάλογα με την νομοθεσία της και ανάλογα με την πολιτική νοτροπία που επικρατεί εκεί, να αποφασίσει όσο γίνεται καλύτερα για το τι θα κάνει. Η δυνατότητα του να υπογράφει ένας πολίτης μια πρωτοβουλία, όντως πρέπει να είναι δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών. Όπως λέει και ο τίτλος της πρωτοβουλίας αυτής. Είναι πρωτοβουλία πολιτών. Άρα πρέπει να έχουν δικαίωμα να υπογράφουν και να υποβάλουν τέτοια πρωτοβουλία Ευρωπαίοι πολίτες. Τώρα για το όριο των κρατών μελών, πόσα πρέπει να είναι. Και εδώ πρέπει να αναρωτηθούμε κάπως. Η πρωτοβουλία αυτή των πολιτών πρέπει να επιτρέπει να γίνεται μια συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό ίσω ο αριθμό των χωρών μελών πρέπει να αυξηθεί. Να λέμε ας πούμε το 1 τέταρτο των χωρών μελών. Γιατί τότε θα έλεγα ότι τότε μόνο μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα γίνεται μια συζήτηση σε πραγματικά ευρωπαϊκό επίπεδο και θα αφορά δηλαδή πολλές χώρες. Τέλος, το θέμα του αποδεκτού μια τέτοια πρωτοβουλίας. Αναρωτιέμαι, η Επιτροπή μας δεν θα έπρεπε να δει κατά πόσο η Κομισιόν από μόνη της πρέπει να αποφασίζει για το αποδεκτό ή όχι μιας πρωτοβουλίας Ευρωπαίων πολιτών. Γιατί τότε η Επιτροπή δεν μπορεί να είναι και αυτή που κρίνει και αυτή που κρίνεται. Δεν μπορεί εκείνη να αποφασίζει για το κατά πόσο είναι αποδεκτή μία ή άλλη ε, πρωτοβουλία, μήπως τελικά θα οδηγηθεί και από κριτήρια πολιτικά και όχι μόνο νομικά. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει και εμείς να βοηθάμε την Επιτροπή στο έργο της, δηλαδή να μην είναι η μόνη που θα κρίνει το αποδεκτό. Να υπάρχει κάποιος άλλος. Είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε το Συμβούλιο, δεν ξέρω, μια που είμαστε συνομοθέτες και δύο οι εμπειρογνώμονες, ειδικοί, πανεπιστημιακοί, νομικοί, δεν ξέρω, κάποιος άλλος πάντως να υποστηρίζει σε αυτό το έργο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην είναι μόνη της που θα κρίνει και θα κρίνεται τελικά. Ευχαριστούμε. Νόκα. Ευχαριστώ, λέει κύριε Τζανόκα. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στους εισηγητές. Συμφωνώ με τις περισσότερες προτάσεις, εκτός από μία θα σας πω μετά. Στηρίζω όμως απόλυτα αυτά που είπατε για το ποιος μπορεί να υπογράψει μια τέτοια πρωτοβουλία. Και ο κύριος Μπάσουλ και οι συνάδελφοι εδώ συμφώνησαν. Αν θέλουμε να είμαστε συνεκτικοί με το έργο μας, πρέπει να τηρούμε τις αρχές μας. Μην ξεχνάτε την έκθεση όλα κάτι που αναφερόταν στην ε, Ευρωπαϊκή Θαγένεια και εγκρίθηκε στην προηγούμενη θητεία. Είχε προταθεί να διευρυνθεί ε, το πεδίο αυτών που μπορούν να ψηφίσουν για τις ευρωεκλογέ. Αν ήταν μόνιμοι κάτοικοι. Και υπάρχει ειδική κατηγορία μονίμων κατοίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είναι όμως πολίτες καμίας ευρωπαϊκής χώρας. Υπάρχει τέτοια περίπτωση και στη Λετωνία, την Εσθονία, και τη Σλοβαδία που είναι απάτριδες ουσιαστικά. Σε άλλη έκθεση και εξετάστηκε και εδώ στην Επιτροπή αυτή η έκθεση Ντερόσα τον Απρίλιο πέρυσι προτάθηκε και οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να συμμετέχουν στις ευρωεκλογέ και στις τοπικές εκλογές. Μία από τις ίδιες τις πρωτοβουλίες στο κάτω-κάτω θα μπορούσε να ήταν μία που έχει να κάνει με αυτό το ζήτημα. Δηλαδή ποιοι μπορούν, ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου στις ευρωπαϊκές εκλογές και να ζητήσουν να βελτιωθεί αυτή η διάταξη για να μπορούν περισσότεροι να ψηφίζουν για τις ευρωεκλογές. Λέω, μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μιας πρωτοβουλίας Ευρωπαίων πολιτών. Εγώ, για παράδειγμα, ευχαρίστω ε, θα ξεκινούσα να υποβάλω μια τέτοια πρωτοβουλία πολιτών. Τώρα, πόσε υπογραφέ χρειάζονται από την κάθε χώρα. Κοιτάξτε, πολλέ πρωτοβουλίε μπορεί να έχουν περιφερειακό χαρακτήρα και μπορεί να έχουν να κάνουν με μικρέ χώρε μέλη. Πάντα. Γιατί το αγωγό, το βαλτικό. Πρόκειται για την βαλτική περιοχή, για μικρές χώρες, τρεις μικρές βαλτικές χώρες. Αν υπάρχει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, οι υπογραφές πρέπει να έρχονται και από μια άλλη μεγάλη χώρα. Ναι, αλλά σε τι αναλογία δεν ξέρω, εδώ δεν συμφωνώ. Αναλογικότητα με τον αριθμό των κατοίκων. Ευχαριστούμε που τηρήσετε το χρόνο σας, η κυρία Ντεμπρούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και συγχαίρω τους συναδέλφους Χόλες και Χέφνερ. Πρέπει η προσέγγιση να είναι πάρα πολύ ανοιχτή, η διαδικασία υποβολής της πρωτοβουλίας της των πολιτών να είναι όσο δυνατόν πιο προσβάσιμη όσο γίνεται και θα χρησιμοποιηθεί από τους πολίτες. Πρέπει λοιπόν να έχουμε τους λιγότερους δυνατούς περιορισμούς που θα τους αποτρέψει, ώστε να μην τους αποτρέψει να προωθήσουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Για τη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση δεν με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη. Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό πολύ σημαντικό εργαλείο για τους πολίτες και χρειαζόμαστε χρόνο για να το φτιάξουμε σωστά. να μην δημιουργήσουμε εμπόδια στη συλλογή των, υπογραφών. Όλε οι πρωτοβουλίε θα είναι, πρέπει να είναι αποδεκτέ σε ψημή που δεν ε, παραβιάζουν βασικέ αρχέ ασφαλεία. Αυτοί που υπογράφουν να είναι οι ίδιοι με τους αναφερόμενους, δηλαδή οποιοδήποτε πολίτης ή κάτοικος της Ένωσης και οποιοδήποτε περιορισμός που θα υποβληθεί αυτόνομα, αυτόματα απαιτεί γραφειοκρατία που θα ελέγξει κατά πόσον υπάρχει περιορισμός, ε, ε, τηρήθηκε ή όχι. Και αυτό είναι άλλος κίνδυνος. Ποιος μπορεί να υπογράφει να είναι μια ανοιχτή διαδικασία γιατί αλλιώ υπάρχει κίνδυνος άγγισης μεταχείριση. Το σημαντικό είναι ένα εκατομμύριο υπογραφές παραπάνω από ένα κράτη-μέλη, ορισμένα κράτη-μέλη, ορισμένο αριθμό, όχι περιορισμοί ούτε στον αριθμό των κρατών μελών, όχι πάρα πολλά, ούτε πάρα πολλέ υπογραφέ από μία συγκεκριμένη χώρα. Πιστεύω ολόψυχα ότι ένα εκατομμύριο υπογραφέ θα πρέπει να αποτελεί υποχρέωση δράσης για την Κομισιόν. Κολάρσκα. Στα αγγλικά ευχαριστώ. Συμφωνώ με τον κύριο Μπουσουτήλ για τον αριθμό ε, προκειμένου να γίνει αποδεκτή. Μπορεί είναι, είναι μικρό το νούμερο αυτό που προτείνεται. Δεύτερον, και ευχαριστώ τους συζητητές για το κείμενό τους. Πώς θα πληροφορήσουμε τους πολίτες για τη νέα αυτή πρωτοβουλία. Χρειάζεται ειδική προσπάθεια για να κυκλοφορήσει αυτή η πληροφορία. Και θα πρέπει η Κομισιόν να δώσει χρήματα και χρόνο για να το πετύχει αυτό. Είναι νέο εργαλείο που θα μας συνδέει με τους πολίτες Τρίτο, για την Επιτροπή μας. Πρώτον, εδώ θα πρέπει να έρχονται οι αναφορές οι οποίες έχουν απορριφθεί κάπου αλλού. Δηλαδή, η, η Κομισιόν, ας πούμε, μπορεί να πει ότι δεν είναι αποδεκτό, δεν πρέπει να συζητηθεί. Πρέπει να υπάρχει ένας άλλος χώρος όπου αυτοί που οργανώνουν την αναφορά να μπορούν να απευθυνθούν και να πούνε βοηθήστε μας δεν συμφωνούμε με την Κομισιόν. Θα μπορούσε η Επιτροπή μας να παίξει αυτό το ρόλο. Θα υπάρξουν πρωτοβουλίες με πάνω από ένα εκατομμύριο επιγραφές συγγνώμη, που δεν θα έχουν ένα εκατομμύριο υπογραφέ, αλλά έχουν να είναι σημαντικέ. Θα μπορούσαμε να τι συζητήσουμε στην Επιτροπή μα. Τι μπορούμε να κάνουμε με αυτές. Είναι ένα σημαντικό σινιάλο από τους πολίτες. Δεν είχαν αρκετή δύναμη να φτάσουν το όριο των υπογραφών. Αλλά θα πρέπει κάπως να το φροντίσουμε. Νταφ. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Ποζωτήλ ζήτησε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων. Εγώ είμαι συνταγματολόγος. και εισηγητής για την ηλεκτρονική μεταρρύθμιση στο Κοινοβούλιο. Συγγνώμη, για την για το εκλογική μεταρρύθμιση στο Κοινοβούλιο. Εγώ θα αναφερθώ μόνο σε ένα σημείο. που εγώ και άλλοι συνάδελφοι στην Συνταγματική Επιτροπή αισθανόμαστε δυσφορία. Ο έλεγχος του αποδεκτού ή όχι, είτε στην αρχή είτε κάπου καθοδόν. Το να υποχρεώσουμε την Κομισιόν να πάρει θέση για το αποδεκτό νημί φέρνει την Κομισιόν σε μια θέση όπου θα είναι και δικαστής και ένορκος. Δεν είναι σωστό αυτό για την Κομισιόν. Είναι ανάγκη να υπάρχει έλεγχος του αποδεκτού. Αν ο κανονισμός συνταχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε με σαφήνεια να λέει ότι οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις αξίες, στόχους και αρμοδιότητες της Ένωσης και να σέβονται τις εξουσίες της Κομισιόν. Όλα αυτά ορίζονται στη συνθήκη της Σαββόνας. Αυτό αρκεί για τον υπεύθυνο πολίτη να το καταλάβει και να το τηρήσει. Είναι ένα σοβαρό συνταγματικό θέμα το οποίο πρέπει να θέσουμε και να απαντήσουμε. Το νομοσχέδιο οποίο ο συνάδελφο ε, Ντάφ επεσήμανε τι κοινέ εργασίε με την Συνταγματική Επιτροπή. Σα λέω κάτι που σκόπευα να πω στο τέλο. Προβλέπονται κοινέ συνεδριάσει με την ΑΦΚΟ. Η άλλη επιτροπή ξεκίνησε πριν από εμά. Εμεί χρειάστηκε να πάρουμε την έγκριση, γι' αυτό καθυστερήσαμε. Αυτοί κάνανε τη συζήτηση, Εμεί την κάνουμε τώρα. Το Σεπτέμβριο η συνεδρίαση θα είναι κοινή. Πάντω οι εισηγητέ συνεργάζονται. Η πρόταση Μπουσουτήλ και η πρόταση Νταφ ήδη έχουν πάρει απάντηση στην κοινή αυτή οργάνωση των δύο επιτροπών. 29 Σεπτεμβρίου συνάντησε με τον Επίτροπο Σεύκοβιτς και με την Επιτροπή ΑΦΚΟ. 30 Σεπτεμβρίου η ΑΦΚΟ καλεί τα Εθνικά Κοινοβούλια και θα είμαστε και εμείς παρόντες. Μέσα Οκτωβρίου έκτακτη συνεδρίαση των δύο επιτροπών για το έγγραφο αυτό. Ίδιες προθεσμίες τροπολογία, ίδιες προθεσμίες για την ψηφοφορία και στην Ολομέλεια. Θα είναι ένα κοινό κείμενο, αν και τυπικά θα είναι δύο χωριστά. Τελευταίος ο συνάδελφος Μποσινάρου. Πολύ σύντομα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτον, Κατά την άποψή μου και ε, κοινώντας το, κοιτώντας το πνεύμα των έπνευστων ε, αυτής της πρωτοβουλίας, η πρωτοβουλία δεν έχει στόχο να δημιουργηθούν νέα πολιτικά εργαλεία, να γίνει πολιτικός ε, θόρυβος, ε, ντόρος ή να λαϊκίσει, αλλά για να αλλάξει ε, να πιέσει το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα ε, που μπορεί ακόμα να εμφανίζουν απροθυμία αυτά τα δύο θεσμικά όργανα. Γιατί έχει άλλο ειδικό βάρος να έχει πίσω σου ένα εκατομμύριο Ευρωπαίους πολίτες. Και να είναι σχεδιασμένη έτσι η πρωτοβουλία ε, ώστε να έχει αποτέλεσμα. Αυτό τι σημαίνει κατά την άποψή μου. Πρώτον, να έχει έτσι ένα σεβαστό αριθμό υπογραφών, εντάξει αυτό, είναι ρυθμισμένο. Ε, σημαντικό αριθμό κρατών μελών επίσης, διότι κάποιοι συνάδελφοι προηγουμένω είπαν ότι δεν μπορεί να είναι πολύ ε, πολύ από λίγα κράτη-μέλη που να σηκωθούν και να γεννούν αυτά ανησυχίε σε άλλα κράτη-μέλη. Α μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ευρωπαϊκές πολιτικές και όχι ξέρω για περιφερειακές πολιτικές ή τοπικά προβλήματα. για τους πολίτες που έχουν δικαίωμα να υπογράφουν μια πρωτοβουλία ε, και οι ίδιοι που έχουν δικαίωμα να κάνουν αναφορά να έχουν και δικαίωμα πρωτοβουλίας. Και ποιος το ελέγχει αυτό, τα κράτη-μέλη. Στα κείμενα που λάβαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Συμβούλιο λέει τα κράτη-μέλη. Και πιθανότατα αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ να είναι να έχουμε ένα τυχαίο έλεγχο αντίστοιχο κάθε 10, 20, 50, δεν ξέρω, αλλά σε όλα τα κράτη-μέλη. Να μην υπάρχουν ε, διαφορετικές προδιαγραφές. Τελευταίο σχόλιο, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα για να συζητήσουμε για τροπολογίες. Θέλω να καλωσορίσω ε, τη συνεισφορά των εισηγητών και να τους συγχαρώ γι' αυτό. Χρειαζόμαστε ευρεία πολιτική στήριξη και εδώ στην Επιτροπή Αναφορών και στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων αλλά και στην Ολομέλεια μετά για να ψηφίσουμε αν όχι ομόφωνα με πολύ μεγάλη πλειοψηφία και μετά να διαπραγματευτούμε το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να φτιάξουμε το καλύτερο δυνατό έγγραφο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνάδελφος ευχαριστώ. σύντομα παρακαλώ. Γιατί έχουμε δυσκολίες. Το Σεπτέμβριο θα το ξαναπούμε. Äh, Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι δύσκολο αυτό αλλά και ωραίο. Γιατί κάναμε ευρύτατη ανταλλαγή απόψεων, ακούστηκαν πολλά θέματα από πολλούς συναδέλφους και τώρα εγώ δεν μπορώ να συνοψίσω και να ε, αναφερθώ εκτενώς σε όλους. Πολύ σύντομα, κάπου που μπορώ να πω ήδη από τώρα κάτι, θα το πω. Πάντως να ξέρετε ότι ε, τις ιδέες σας θα τις ε, εξετάσουμε πάρα πολύ σοβαρά και θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ κύριε Βαλένσα. Νομίζω δεν χρειάζεται να αντιδράσω άμεσα. Ο κύριος Μπούσου έφερε εδώ ένα ολόκληρο φάσμα, ένα μπουκέτο θεμάτων. Ε, κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων σας απάντησαν σε αυτό. Και επίσης τα έγγραφα Λαμασούρ και ή θα σας τα στείλουμε ευχαρίστω και σε όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής μας. Αυτό ισχύει και για το σχέδιο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, τη θέση του Συμβουλίου. Γιατί μου ζήτησαν κάποιοι συνάδελφοι ότι θα τα ήθελαν αυτά και δεν τα έχουν. Μπορούμε να τα στείλουμε έτσι συνολικά. Λέει, θα σας φαίνεται πολύ λίγος αριθμός ε, ε, το 7 για τους αρχικούς ε, υπογράφοντες. Στην πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα πρόσωπο, ξέρετε, και στην πρώτη Συμβουλίου. Και εμεί ανησυχούμε γι' αυτό το ένα. Ιδιαίτερα στη διαδικασία την διαδικτυακή πολύ γρήγορα γράφει κάποιος κάτι στον υπολογιστή του και ξεκινάει την πρωτοβουλία. Το βαφτίζει πρωτοβουλία των πολιτών. Όχι, εμείς είπαμε ε, να είναι μερικοί ήδη που να έχουν σκεφτεί, να έχουν συζητήσει αυτό το θέμα, να το έχουν επεξεργαστεί και να είναι και μια δημοκρατική δομή. Δηλαδή να γνωρίζουμε ποιος έχει ε, δικαίωμα, ποιος αιτιολογείται και δικαιολογείται να συζητάει για αυτή την πρωτοβουλία. Γι' αυτό προτείναμε το 7. Χαίρομαι που λέτε ότι πρέπει να είναι περισσότεροι, αλλά είναι νέα ιδέα. Ε, εμείς τώρα τη φέραμε στο παιχνίδι για να δώσουμε μεγαλύτερο κύρος για το αποδεκτό ή μη. Νομίζω ότι είναι σαφείς οι κανόνες εδώ. Θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μάλλον να μην αντιτίθεται στο άρθρο 6 της Σύνδεξης της Αβώνας και του Θεμελιώδου Χάρτη ε, ούτε λοιπόν στις αξίες και τις αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί που δυσκολεύουν τα πράγματα είναι στα παραδείγματα που δίνεται. Γιατί ο καθένας από εμά έχει στο μυαλό του αμέσως παραδείγματα που θα του άρεσαν τέτοιες πρωτοβουλίες και κάποια άλλα που δεν θα του άρεσαν. Αλλά δεν μπορεί να είναι αυτό ο γνώμονας. Ο γνώμονας θα είναι να ανοίξουμε το δρόμο για τους πολίτες. Έχουμε πολλά προηγούμενα ακούσαμε και προηγουμένω εκπρόσωποι τη βιομηχανία, ομάδε πίεση κτλ. απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για πρώτη φορά τώρα ανοίγει ένα δρόμο για να μπορούν να απευθύνονται οι πολίτε με οργανωμένο τρόπο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και είναι ένα είδο γλώσσα των πολιτών, εγκαθίδρυση ενό διαλόγου στην Ένωση με του πολίτε. Είμαι και εγώ πεπισμένος, όπως και η Νταγιάννα Γόλης, ότι με το διάλογο, τη συζήτηση, τελικά θα προχωρήσει η Ευρώπη. Αυτό δεν θέλει λοιπόν να βλάψει την Ευρώπη. Να σας πω κάτι, στη Γερμανία έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα πρόσφατα που λέγει ότι ακόμα και οι κριτικές συζητήσεις κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης από επικριτές και αντιπάλους της τελικά εξυπηρέτησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί οι πολίτες προβληματίστηκαν, ενημερώθηκαν και έλαβαν θέση και τελικά είναι υπέρ της Ευρώπης και όχι εναντίον της ακόμα και μια κακοπροαίρετη ας πούμε. Και η λήψη των αποφάσεων εδώ δεν είναι των πολιτών. Απλώς οι πολίτες ε, αποτείνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάνουν προτάσεις και τα αρμόδια θεσμικά όργανα έχουν τη διακριτική ευχαίρεια να τα δεχθούν ή όχι. Όπως με το δικαίωμα ε, για τις αναφορές. Γιατί να μην έχει το δικαίωμα ο καθένας που έχει δικαίωμα σε αναφορά να κάνει πρωτοβουλία θα ήταν τελείως διαφορετικά εάν ε, πρόκειται για εκλογές ή για αποφάσεις. Εδώ πρόκειται για προτάσεις και μόνο, γι' αυτό έχουμε λάβει αυτή τη θέση. Αλλά αν θέλετε να το συζητήσουμε και στη συνέχεια. Για τους 18 μήνες, τώρα πρέπει να σας πω... Εσείς λέτε ότι είναι μεγάλο χρονικό διάστημα υπερβολικά. Μα κοιτάξτε, συζητάμε για ένα εργαλείο πρωτόγνωρο, δεν υπήρξε στο παρελθόν. Σε 23 διαφορετικές γλώσσες, 27 διαφορετικά κράτη να ε, οργανώνεται συλλογή υπογραφών. Ήδη έχουμε πολλές πρωτοβουλίες που προσπάθησαν να το κάνουν με ε, τις συνθήκες της Αβώνας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σκεφτείτε και ε, όταν θα έχει αποφασίσει για το αποδεκτό Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να τυπώσουν το υλικό, να το οργανώσουν στις χώρες να βγει ο κόσμος να μαζεύει υπογραφές. Δεν θέλουμε μόνο online. Εντάξει, στο διαδίκτυο είναι πιο γρήγορα. Αλλά ε, στο δρόμο είναι ε, περισσότερα τα τεκτενόμενα γίνεται συζήτηση. Δεν πατάς ένα κουμπί σε ένα κομπιούτερ, οπότε χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Και το τελευταίο σε σχέση με αυτό που είπατε, δεν θα πρέπει να ορίσουμε από τώρα εμείς το τι θα συμβεί μετά. Πρέπει να σας πω για όλους τους συζητητές ότι αυτό είναι ακριβώς το αποφασιστικό για μας, διότι έχουμε δικαίωμα αναφοράς και εδώ πρόκειται για ένα νέο δικαίωμα, περισσότερο. Και ερώτηση, γιατί να ε, μαζέψουν ένα εκατομμύριο ε, υπογραφές οι πολίτες. Αυτό είναι τεράστια ενέργεια και ανθρώπου ώρες ε, ε, αφιερώνεται εκεί και χρόνος και ενέργεια και τελικά να πέσει αυτό στο κενό. Νομίζω ότι μια ακρόαση των ε, διοργανωτών και αιτιολογημένη απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή να τεκμηριώνει για την απόφαση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι το ελάχιστο που θα πρέπει να επιφυλάσσεται στους πολίτες για να μην δημιουργήσουμε ένα όργανο που θα ενισχύσει την απογοήτευση ε, και να μην αποκαρδιώνει τους πολίτες, αλλά να τους ευθαρρύνει. Το τι θα γίνει μετά είναι για μας αποφασιστικό και στη συνέχεια των συζητήσεων μας σίγουρα θα μας απασχολήσει. Για την κυρία Λεγκρίπ. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το ζήτημα. Εάν θα πρέπει να αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ε, δεν μπορεί να είναι κριτής και κρινόμενος. Ε, πολύ ενδιαφέρουσες ε, ιδέες αλλά και προβληματικές από τη φύση τους και πάλι. Θα μας απασχολήσει στο μέλλον, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες αυτό, γιατί η Τατιάνα Ζανόκα, το θέμα της εθνικότητας και της ιδιότητας του πολίτη είναι πολύ σημαντικό δεν θέλω να επιμείνω γιατί μου κάνει νοήματα η πρόεδρος. Αυτό το θέμα των μικρών κρατών είναι μια δυσκολία που γράφεται και στη συνθήκη της Λισαβόνας την ίδια. Το λέω ξεκάθαρα γιατί είχαμε διαπραγματευτεί και εγώ υποστήριζα μια άλλη πρωτοβουλία των πολιτών απέναντι στην τακτική συνέλευση, τα διαφορετική αρχική διατύπωση. Αλλά στην τωρινή διατύπωση όντως ένα εκατομμύριο υπογραφέ είναι που πούμε, για τις χώρες φαλτικής και μόνο παράδειγμα και μετά σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχει η ρητή επιθυμία να μην είναι απλώ και μόνο περιφερειακή διαταξή. Η σταδιακή αναλογικότητα απορρέει εμπειρικά από τη συλλογή των, εμπειριών, των, υπογραφών. Τώρα δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, απλώς να τα έχετε υπόψη σας αυτά για τη συνέχεια της συζήτησης. Για την κυρία Ντεμπρά συμφωνώ πάρα πολύ. Δεν θα πρέπει να είμαστε υπερβολικά περιοριστικοί και να δεσμευτούμε η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή να αντιδράσει. Κυρία Κολάσκα Μπαμπίνσκα, ναι, οπωσδήποτε έχετε δίκιο να δημοσιοποιηθούν όλα αυτά. Είναι σημαντικό στόχος μας και θα πρέπει πολύ συγκεκριμένα να πούμε στου πολίτε ποιε θα είναι οι κατευθυντήριε γραμμέ. και σε σχέση με το δικαίωμα αναφορά Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να παίξει μεγάλο ρόλο εδώ και να δούμε και ποιο όργανο του Κοινοβουλίου ε, είναι αρμόδιο, ποιο άλλο όργανο του Κοινοβουλίου έχει τόση εμπειρία και τόση εξοικείωση σε θέματα πολιτών από την Επιτροπή Αναφορών. Και μετά, ποιο ελέγχει και αν χρειαζόμαστε κανένα τέτοιο έλεγχο. Ενδιαφέρον και αυτό, θα το σημειώσουμε. και αυτά που είπε ο Βίκτορ Μποστινάρου επίσης για την προοδευτική, προοδευτικά μειούμενη αναλογικότητα. Δεν έχουμε χρόνο τώρα να σας τα εξηγήσω επί της ουσίας, αλλά θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να τα κουβεντιάσουμε. Ήταν η πρώτη ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μετά από μερικά λεφτά δεν θα έχουμε διερμηνίες. Θα συνεχίσουμε στα αγγλικά αν θέλετε πολύ σύντομα στο λόγο ο Σνάφου Γκέριγκερ για το σημείο 12 13 Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λυπάμαι για το ότι έχουμε μόνο δύο λεπτά για να συζητήσουμε ένα τόσο σημαντικό θέμα. και δεν συμβαίνει αυτό πρώτη φορά. Πώς είναι δυνατόν να εξηγήσω τη θέση της Κομισιόν και να συζητήσουμε κιόλας τα δύο λεπτά που μας μένουν καλύτερα να τα αφιερώσουμε σε κάτι άλλο να συζητήσουμε το θέμα αυτό το απόγευμα σοβαρά Πρόεδρος. Συμφωνώ. Ωραία. Ας πάμε το απόγευμα. Με το βάλουμε πρώτο το Σεπτέμβριο το απόγευμα το Σεπτέμβριο. Do you want to vote for this proposal? September. September. θα πρέπει να αναβληθεί και το επόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη. Είναι παρόν όμως ο κύριος Κλάιν. Μπορείτε να έρθετε στις 3 για να το αναπάρουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι. Βεβαίω, μπορώ... So θα ακούσουμε μόνο την Επιτροπή γιατί δεν μπορεί να είναι εδώ το απόγευμα, λέει. Miss Minor cannot come in the afternoon. Okay. Δεν μπορεί, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να παραστεί το απόγευμα. Ναι, αλλά έχουμε πολλές ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει η κυρία Τιγκέ. Δεν μπορεί να έρχεται κάποιο χωρί να μα ακούσει τι ερωτήσει μα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι λογικά αυτά τα πράγματα. Συμφωνώ, Πρόεδρο. Αλλά για το άλλο θέμα είναι αυτό, όχι για το δικό σα για τον κύριο Κλάιν. Καλά. Ε, then we were informed he cannot come, but he sends someone. But if δεν μπορεί να έρθει, αλλά θα στείλει κάποιον. Αλλά τώρα μας λένε ότι δεν θα είναι κανένας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να οργανωθεί για να είναι εδώ. Εδώ είμαι, λέει η Επιτροπή. Δεν κατάλαβα, είναι παρεξήγηση. Μα το αναβάλαμε για το απόγευμα, δεν είπαμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μιλήσει τώρα, διότι η κυρία Μέγερ δεν μπορεί να έρθει το απόγευμα. Αλλά αναβάλαμε το θέμα και θα ακούσουμε τον κύριο Κλάιν και τους υπολείπους το απόγευμα. Χωρίς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στείλει κάποιον άλλον το απόγευμα. Γιατί έχουμε σημαντικές ερωτήσεις να τις κάνουμε. Εγώ δεν θέλω να ακούσω την απάντηση πριν να κάνουμε τις ερωτήσεις μας. <laughs> Yes, I know, but this is the, the situation. We can, we can listen to the answer